Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην ε, συνεδρίασή μας αυτή την εβδομάδα. Ιδιαίτερα βεβαίω θα καλωσορίσω την Επίτροπο, την κυρία Γκέγγεν Κουίν, η οποία θα συζητήσει μαζί μας ναι, αυτό είναι το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Βεβαίως πρώτα απ' όλα έχουμε να διεκπαιρεώσουμε κάποια οργανωτικά. Πρώτα απ' όλα για την ημερήσια διάταξη το σημείο 5 και 6 αλλάζουν σειρά μεταξύ τους. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Το έχουμε συζητήσει. Κατόπιν υπάρχουν τα πρακτικά και εκεί πέρα αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις εγκρίνονται. Σήμερα, κατά εξαίρεση, έχω να πω δύο-τρία πράγματα ως ανακοινώσεις και θα σας παρακαλέσω και όλας να τα μεταφέρετε αυτά στις ομάδες σας και να επανέλθετε. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο είναι πως Ολοκληρώσαμε τον τριμερή διάλογο για το ERP που ήταν δύσκολο. Η κυρία Μπρέντ και κάποιοι συνάδελφοι διαπραγματεύτηκαν. Ήταν δύσκολο να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα με το Συμβούλιο γιατί υπήρχε μία μειοψηφία που μπλόκαρε τα πράγματα αλλά παρόλα αυτά ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις και θέλω να τους συγχαρώ. Ε, δεν είναι εδώ πέρα βεβαίως κρίμα Δεύτερη παρατήρηση στην διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών είχαμε μια συζήτηση στο Στρασβούργο για τις συμφωνίες στην πρώτη ανάγνωση κατά το οποίο και θέλω να σας αναφέρω κάποια αρκετά σημαντικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια αξιολόγηση του σε ποιο μέτρο και σε ποιο βαθμό ε, Λαμβάν χώρα συμφωνεί στην πρώτη ανάγνωση και βεβαίως ε, αυτό συμβαίνει όλο και συχνότερα. Μιλάμε για ένα 70%. Βεβαίως ένα νούμερο δεν είναι αποφασιστικό. Εγώ συμφωνώ με την ανησυχία των προέδρων των ομάδων ότι πρέπει να προσέχουμε να μην ε, διακινδυνεύσει έτσι η δημοκρατική διαδικασία γιατί ο μεμονωμένος βουλευτής δεν έχει πλέον ευκαιρία να παρέμβει, κάτι το οποίο εις βάθος χρόνου δεν είναι καλό. Υπάρχουν βεβαίως κάποιες επιτροπές όπως η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων οι οποίες ε, συμφωνούν σε πάρα πολλά πράγματα, σε πάρα πολλές λεπτομέρειες οι οποίες δεν είναι επίμαχες ε, και βεβαίως εκεί πέρα μπορούμε απλώς να ψηφίζουμε. Οπότε σωστό είναι να υπάρχουν διορθώσεις, να εργαζόμαστε εκ των προτέρων και δεν ξέρω, θα μπορούσε ίσως να μου το υπενθυμίσει η γραμματεία, να γνωρίζουν ε, και τον ε, κανονισμό όλοι οι βουλευτές γιατί εάν μιλάμε για συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση υπάρχει μια ακολουθία που πρέπει να ακολουθεί να γίνουν τα πράγματα σωστά δηλαδή όταν γίνεται κάτι τέτοιο θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία. Γι' αυτό θα ήθελα να το τηρείτε αυτό. Και η τρίτη ανακοίνωση, κάτι το οποίο απασχόλησε και τους συντονιστές, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος υπάρχει μια έκθεση πρωτοβουλίας για την ανακοίνωση της Κομισιόν για τις εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου. Εκεί πέρα είπα πως ε, θέλουμε και εμείς να λάβουμε μέρος σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 51. Δεν είναι δυνατόν ε, να τα κάνει αυτά τα πράγματα τα οποία μας αφορούν οπωσδήποτε αποκλειστικά μόνη της η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είχαμε ήδη κάποια προβλήματα. Εγώ ανέφερα την 51, το απορρίπτει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρέπει να δούμε τώρα πώς θα προχωρήσουμε συναντήθηκα με τον Γιώ Λάινεν, τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και αυτός προτείνει να, να ακολουθήσουμε το άρθρο 50. Είπα να το συζητήσουμε εάν διασφαλιστεί σε ποιους τομείς είμαστε μετά αρμόδιοι. Πρέπει να οριστεί δηλαδή επακριβώς ε, π.χ. στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οτιδήποτε αφορά βιομηχανία, έρευνα ενέργεια. Όλα αυτά είναι αποκλειστική δική μας αρμοδιότητα. Η γραμματεία τώρα ζήτησε από τη γραμματεία να αναφέρει ποιοι είναι οι δικοί μας τομείς ε, αρμοδιότητες. Θα τα αποστείλω αυτά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και θα παρακαλέσω να συμφωνήσουμε σε αυτά. Ε, Βεβαίω είμαστε διατεθειμένοι για συμβασμό μόνο, μόνο τότε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να διαπραγματευόμαστε τα τρία τέταρτα των ε, θεμάτων αυτών που μας να φορούν. Εντάξει, μία φορά πέρασε έτσι, αλλά τώρα πρέπει να το δούμε κάπως πιο εντατικά. Αυτή ήταν η τρίτη και τελευταία ανακοίνωση. Θα σας ακούσω τώρα. Α, συνεχά και τον κύριο Φανμπρέν, ο οποίος τώρα είναι εδώ πέρα και τα ακούει. Νομίζω ολοκληρώσα τι ανακοινώσει με αυτά και αν δεν έχετε εσείς ε, τίποτα άλλο να προσθέσετε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4 τη ημερήσια διάταξη στην επίσκεψη και στην συζήτηση βεβαίως ε, με την κυρία Γιώργεν Κουίν. Επιτρόπου για την έρευνα, καινοτομία και επιστήμη και η πρότασή μου είναι να κάνετε μία σύντομη δήλωση, μετά να δεχτείτε ερωτήσεις. Θα κοιτάω και εγώ τον χρόνο και μετά θα δώσει και απαντήσεις η κυρία Επιτροπός. Λοιπόν, καλώς ήρθατε κύριε Επιτροπέ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, ευκαιρία που μου δώσατε να συναντηθούμε σήμερα το απόγευμα και να παρουσιάσω το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011 σχετικά με την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη και να παρουσιάσω και την ε, πρωτοπόρο καινοτομία μας ε, η οποία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Οκτωβρίου για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την φόρο ανάπτυξη πρέπει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της κοινωνίας και ε, να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη επίπτωση των ε, χρηματοδοτήσεών μας με περισσότερη καινοτομία. Θα επανέλθω στα θέματα αυτά αργότερα. Απλώς η εφαρμογή θα πρέπει να ε, είναι κάτι που θα έχουμε υπόψη μας σε συνδυασμό με το σχεδιασμό για να επιτύχουμε τον στόχο μας στο 2014 σχετικά με την έρευνα και να δημιουργήσουμε ένα νέο πρόγραμμα. Παραμένουν όμως πολλά ερωτήματα για το πώς το πρόγραμμα πλαίσιο 8 θα διαρθρωθεί και πώς θα εξυπηρετήσουμε τους στόχους της στρατηγικής του 2020 και την καινοτόμα ένωση όσο δυνατόν καλύτερα. Οι εμπλεκόμενοι επόμενοι ε, θα ερωτηθούν προτού Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήξει στις προτάσεις της και αυτή η διαβούλευση θα βασιστεί σε μια ανακοίνωση που θα αναφέρεται στα βασικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν για το 2011 και η υιοθέτηση του προγράμματος και των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο έχει προβλεφθεί για το έτος του 2011. Δεδομένου ότι η πρόοδος είναι αργή, θα πρέπει να προτείνουμε για το 2012 ένα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη το οποίο θα καταλύει τα εμπόδια στην κινητικότητα και στην διασυνοριακή συνεργασία για να μπορέσει να, τους επιτύχει, να την εφαρμογή του το 2014. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε επίσης μία συνέργεια με το νέο πρόγραμμα πλαίσιο και ε, με τις άλλες πρωτοβουλίες που είναι η ψηφιακή ατζέντα, η ε, νεότης εγκινήση, η ε, βιομηχανική πολιτική και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και εργασιών. Το πλαίσιο αυτό είναι ένα φιλόδοξο πρώτο βήμα για να αναπτυχθεί η πρότασή μας και να μπορέσει μετά από τη διαβούλευση το 2011 να παρουσιαστεί σαν πρόταση πλαίσιο το 2012. Θα προτείνουμε μία πρωτοβουλία η οποία να ανταποκρίνεται στην την στρατηγική του 2020 και θα μπορέσει να επιτύχει την βιολογική οικονομία μέχρι το 2020 ε, εμπλέκοντας και τη βιομηχανική και την γεωργική βιολογική οικονομία. Θέλω όμως τώρα να σας πω ποια είναι η πιο βασική μας πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχω περιβάλει όλα τα στοιχεία τα οποία περιέχει και ε, πολλά από τα σχόλια τα οποία έλαβα αναφέρονται στα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία του οικολογικού συστήματος καινοτομίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βασιζόμαστε σε δέκα στοιχεία κλειδιά. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει μέτρα για να βελτιώσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, να προωθήσει τη χρηματοδότηση στηριακή μορφή η οποία θα μοιράζεται τον κίνδυνο και ε, να ταυτίσει τις ε, καινοτόμες επιχειρήσεις με ε, επιχειρηματίες και επενδυτές. Επίσης θα επιταχύνουμε τις ισχύουσες ερευνητικές πρωτοβουλίες και θα μπορούν να μεταφερθούν και και ε, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα κατά τρόπον ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ε, πρόσβαση ή στην έρευνα η οποία χρηματοδοτείται από το δημόσιο. Υπάρχει ήδη ε, συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας που θα ενισχυθεί. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταρτήσει ένα ε, Συμβούλιο Ευρωπαϊκού Σχεδίου και ε, Αριστείας ε, με την ανάλογη σήμανση. Τέταρτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταρτήσει ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα με βαθμολόγηση κατά τρόπον ώστε να προτείνει την καινοτομία σαν σημείο το οποίο θα εστιάζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η Επιτροπή Πέμπτων θα προτείνει στις κυβερνήσεις να καταρτήσουν προϋπολογισμούς για τις δημόσιες προμήθειες καινοτόμων προϊόντων και ε, υπηρεσιών κατά τρόπον ώστε να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των διαφόρων διαφόρων κρατών μελών. Έκτον, η Επιτροπή θα καταρτήσει μία νομοθετική πρόταση που θα επιταχύνει τα ε, ήδη ισχύοντα. Έβδομα, η ε, πνευματική ιδιοκτησία της Ευρώπης και το σύστημά της πρέπει να ενισχυθεί για να εξοικονομήσουμε 250 εκατομμύρια το χρόνο μέσω του, της συμφωνίας για το σύστημα διπλωμάτων ευρασιτεχνίας. Ογδόν θα υπάρχει διαρθρωτική χρηματοδότηση και βοήθεια για να προωθηθεί η καινοτομία μέσω των διαρθρωτικών προγραμμάτων καινοτομίας από το 2007 μέχρι το 2013. Θα προτείνουμε ένα πρόγραμμα πλαίσιο το οποίο θα εστιάζεται περισσότερο στην καινοτομία και το 2011 θα αναθεωρήσουμε το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. 9. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκεντρώσει 25 δείκτες για την βαθμολόγηση αποδόσεως στην έρευνα και στην καινοτομία βασιζόμενοι στις ε, αναπτυσσόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν καλύτερα στην οικονομία τα επόμενα δύο χρόνια. Δέκατον, ε, θα υπάρξει ευρωπαϊκή συνεργασία καινοτόμα η οποία θα κινητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους και θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να ηγηθεί. Οι συνεργασίες αυτές θα ε, επιταχύνουν την έρευνα και την ανάπτυξη, θα συντονίσουν τις επενδύσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, προσελκύσει ε, χρηματοδότηση, ένα πιλωτικό πρόγραμμα συνεργασίας θα προωθηθεί το 2011 για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για πρώτες ύλες μη ενεργειακές και για η φόρα και παραγωγική γεωργία. Θέλω να σας διασφαλίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη για να διερευνήσει δυνατότητες, δυνατότητες συνεργασίας καθώς επίσης και ε, την ε, διαχείριση και τη δομή αυτών των συνεργασιών η πρωτοβουλία αυτή συζητήθηκε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 12 Οκτωβρίου και ε, θα παρουσιαστεί στο επόμενο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 26 Νοεμβρίου και ο πρόεδρος Μπαρόζο θα το παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Θα ήθελα πολύ να γνωρίζω τις απόψεις σας σχετικά με το θέμα αυτό. Ξέρω ότι η κυρία Τζούντιθ Μέρκης ε, είναι η για αυτό το, αυτή την έκθεση για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο δίκαια και πιο πράσινη κοινωνία και είμαι βέβαιος ότι ο, πρόεδρος Μπαρόζο θα στηριχτεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι θα υλοποιήσει την η Ευρωπαϊκή Ένωση με ανακαινήσεις. Ευχαριστώ. Έχω ήδη τους πρώτους ομιλητές και δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, εξ ονόματος της ομάδας μου και προσωπικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Θα είμαι πολύ σύντομη, θα υποβάλω δύο ερωτήσεις. Μία ερώτηση και θα ήθελα να υποβάλω και ένα σχόλιο. Κατά την άποψή μας, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και όπως ελέγχθη εδώ, προγενέστερα, όταν βρεθήκατε εδώ μαζί μας ή απαντώντας σε γραπτές ερωτήσεις βλέπουμε ότι έχουμε τις, τους 25 συντελεστές που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καινοτομία καθώς και την επιτήρηση των πραγματικών καινοτόμων σχεδίων. Αυτό αποτελεί μία πρόθεση του θέματος που είναι ύψης της σημασίας. Ως προς την εξέλιξη του προγράμματος ITER και την χρηματοδότησή του, όπως ξέρετε κυρία Επίτροπε, η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σε σχέση με την εξέλιξη του προγράμματος ITER είπε ότι θα αυξηθούν οι δαπάνες κατά 2, από 2,7 σε 3,5 εκατομμύρια. Μετά όμως το Συμβούλιο μείωσε αυτό το ποσό σε 6.700.000 ε, μεταξύ του 2012 και 2020. Μιλάμε για μια αύξηση της γραμμής 1α μέσα στα πλαίσια του 7ου προγρα... προγράμματος πλαισίου της τάξης των 470 εκατομμυρίων από πού προέρχεται η χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ. Όπως ξέρετε η γραμμή 1α είναι αρκετά προβληματική γιατί μιλάμε για το πρόγραμμα στρίκτο σένσου και όχι για έργα υποδομών. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο στην παρούσα φάση του ίτερ να χρηματοδοτηθεί από αυτή τη γραμμή, πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την χρηματοδότηση του 7ου προγράμματος δράσης με βάση την προβλεπόμενη ε, χρηματοδότηση, όπως δηλαδή είχε προβλεφθεί αρχικά. Αυτό το σχολιάσαμε πολλές φορές σε αυτή την Επιτροπή και είναι γεγονός ότι θα θέλαμε ορισμένες διευκρινήσεις επί του θέματος. Ε, κυρία Επίτροπε, άκουσα με μεγάλη προσοχή. Αυτά που μας είπατε είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο σημεία. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Πιθανόν από δική μου κακή ενημέρωση δεν έχω καταφέρει μέχρι σήμερα να μάθω τι ακριβώς συνέβη με τη στρατηγική της Λισαβόνας δεν ξέρω κανένα στοιχείο το οποίο να μου λέει πώς τα καταφέραμε ακριβώς με τη στρατηγική αυτή και κατά πώς τώρα έρχεται στο προσκήνιο το όραμα του 2020. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν η στρατηγική της Λισαβόνας έχει εξέλιξη σε αυτό το όραμα του 2020 και σε περίπτωση που όπως οι κακές γλώσσες, γιατί όπως σας είπα στοιχεία εγώ δεν βρήκα, λένε ότι δεν τα πετύχαμε καλά με τη στρατηγική της Λισαβόνας, τι μέτρα έχουν ληφθεί σε αυτό τον προγραμματισμό για το 2020 να, να μην μας ξανασυμβεί κανένα κακό. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι είδα στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο Innovation Union ότι ανάμεσα σε αυτά που ενδιαφέρουν την Επιτροπή και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 7.2 την ενδιαφέρει η ίδρυση, η θέσμηση ενός ε, μοναδικού δίκτυ μέτρησης της καινοτομίας έτσι ώστε να υπάρχει και μια διεθνής συγκρισιμότητα, international comparability. Στην έκθεση αυτή βλέπω ότι η Επιτροπή μας διαβεβαιώνει σύμφωνα με τις ε, εισηγήσει του High Level ε, Panel ότι σε δύο χρόνια θα έχει ανα, αναδειχθεί ένας τέτοιος δείκτης. Η ερώτηση μου είναι, αφού οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Βραζιλία έχουν ήδη αναπτύξει το Star Matrix, το οποίο μετράει ακριβώς αυτό που θέλει να μετρήσουμε κι εμείς, δηλαδή τη σύγκριση των δικτών της καινοτομικότητας, σε σχέση με τα output, σε σχέση με τα εξαγόμενα της innovation, για ποιο λόγο δεν κάνουμε χρήση ή δεν συμβουλευόμαστε αυτόν τον δείκτη που είναι έτοιμος και δεν χρειάζεται να περιμένουμε και δύο χρόνια. Σε ευχαριστώ πολύ. Ford. Thank you very much, Commissioner. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και χαιρόμαστε που ακούμε πως είστε τόσο πολύ άσχολοι κύριε ερωτήσεις Πρώτα απ' όλα για τη χρηματοδότηση του προγράμματος πλαισίου. Ένα πολύ σημαντικό θέμα για την έρευνα και την επιστήμη στη χώρα μου, όπου μου λένε συνεχώς οι ερευνητές πόσο σημαντική είναι η συνεργασία και η κοινοτική χρηματοδότηση για να υπάρξει καινοτομία στην επιστήμη. Συνεργάστηκα με την κυρία Ταβάιο για την απλοποίηση του προγράμματος 7 ε, και θέλω να μάθω πως πώς σκοπεύετε να το εφαρμόσετε ώστε να το πιο γρήγορα. Μία από τις συστάσεις ήταν οι συμμετέχοντες να μπορούν να χρησιμοποιούν τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές και υπάρχει ανησυχία από πολλούς συμμετέχοντες ε, για το κόστος ε, του προσωπικού και εάν ε, θα τους επιτραπεί να χρησιμοποιούν τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές θα αποφευχθεί σύγχυση. Το δεύτερο ερώτημα όταν ε, επανήλθε για μια δεύτερη θητεία ο κύριος Μπαρόσο είπε πόσο μεγάλη σημασία αποδίδει να, υπάρχει, να υπάρχουν επιστημονικές συμβουλές για την Ευρώπη. Τι γίνεται με αυτό, η κυρία Μέρκες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που παρευρεθήκατε εδώ για να μας ε, μιλήσετε για την κατάσταση καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να φτάσουμε στους στόχους μας μέχρι το 2020, όπως είναι γνωστό. Είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό να διασαφηνίσουμε την δομή διακυβέρνησης ε, της εταιρικότητας αυτής. Ε, μπορείτε όμως να μας αποκαλύψετε πώς θα έχει αυτή η διακυβέρνηση, πώς θα συσταθεί. Μιλάμε για ένα νέο μέσο, διότι από όσο διαπιστώνω δεν πρόκειται για ένα νέο μέσο, Πρόκειται για την ανασύσταση ενός ε, παλαιού μέσου. Το οποίο παρουσιάζει μία καθαρά επίπλαστη εικόνα. Αυτό είναι ένα θέμα κλειδί λοιπόν και μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα ορίσουμε την ατζέντα ως προς τις εταιρικές σχέσεις καινοτομίας και πώς θα αναθεωρήσουμε τις ε, ε διάφορες προκλήσεις, τις προκλήσεις μέχρι το 2020, διότι πρόκειται για ένα ρευστό ζήτημα. Ίσως οι προκλήσεις του 2013 είναι διαφορετικές από τις σημερινές και ούτω καθεξής. Ε, ως προς τις οικονομικές εταιρικές σχέσεις, συμφωνώ με τον συνάδελφο Τσουκαλά πώς θα επιτηρήσουμε τα πάντα και πώς θα ενισχύσουμε τα αποτελέσματα των παλαιότερων εταιρικών σχέσεων. Επίσης, ένα ουσιώδες ζήτημα είναι η χρηματοδότηση των εταιρικών αυτών σχέσεων. Μιλήσατε για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν μιλήσατε όμως για το πρόγραμμα καινοτομίας γιατί υπάρχουν χιλιάδες τρόποι χρηματοδότησης της ε, καινοτομίας. Θα ομαδοποιήσει η Ένωση τα πάντα έτσι ώστε να υπάρχει μια πραγματιστική προσέγγιση, διότι η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης σημαίνει και αποτελεσματικότητα της ίδιας ε, της ε, συνολικής χρηματοδότησης και τα πάνω ως προς τη μεταφορά γνώσεων που είναι η πέμπτη ελευθερία μπορείτε να μας πείτε πώς η μεταφορά γνώσεων μπορεί να προαχθεί μέσω καινοτόμων εταιρικών σχέσεων, διότι αυτό έχει σχέση και με τα διπλώματα τεχνίας και με την ενιαία αγορά. Τέλος, μιλήσατε για το πώς μπορούμε να προσελκύσουμε τα ταλέντα. Χρειαζόμαστε Επανεπιστήμια παγκόσμια σε εμβέλειας. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Διότι ε, όπως ξέρουμε ότι όπως ξέρουμε η εκπαίδευση δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πώς συνάδει με την ε, καινοτομία. Uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Επίτροπο, λέει ο κύριος Λάμπερτς, και να την ευχαριστήσω για αυτά τα ενθαρρυντικά λόγια ως προς τους, ως προς τους εταιρικούς στόχους. Πολύ καλή η επιλογή. Αυτή την επιλογή θα έκανα και εγώ. Μιλάτε για ανοιχτή ε, πρόσβαση της έρευνας που χρηματοδοτείται από το δημόσιο. Μιλάμε για IPR για το ERC και EIT και μιλάτε για προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές είναι κρίσιμης σημασίας. Η, η ηλεκτρονική κινητικότητα, για παράδειγμα. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των προδιαγραφών. Ίσως θα μπορούσε να βελτιωθεί κάπως το έγγραφο σε ορισμένα σημεία ως προς την ε, προσέλκυση ταλέντων, αυτό που με ενοχλεί είναι ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μεγάλο απόθεμα ε, νέων ταλέντων. Μιλάμε για το πρόγραμμα Youth on the Move. Έχει σημασία να δούμε και τους μετανάστες ή αυτοί που, οι νέοι που προέρχονται από μία γενεά μεταναστών. Δηλαδή πριν προσελκύσουμε ταλέντα από την αλλοδαπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, τα ταλέντα που διαθέτουμε. Ως προς τις ε, εταιρικέ σχέσεις καινοτομία, η ανησυχία μας είναι ότι δεν πρέπει να επιδοτούμε την βιομηχανία θα πρέπει να υπάρχουν δεσμεύσεις και από τις δύο ή τις τρεις πλευρές. Και εδώ μιλώ και για την χρηματοοικονομική δέσμευση της Ευρώπης. Επίσης, θα προτείνουμε στους συναδέλφους ότι όσον αφορά την ε, χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση θα υπάρξουν μακροοικονομικές ανισορροπίες και θα θέλαμε ο συνάδελφός σας ε, Ρεν να ασχοληθεί και με θέματα αποδοτικότητας της ενέργειας και των πόρων που έχουν άμεσο αντίκτυπο. Άρα, επειδή η Πιλάρ θα ε, ασχοληθεί με το πρόγραμμα ITER, θα ήθελα, κυρία Επίτροπε, να δείτε υπόψη τις δύο σας ιδιότητες. Ήσασταν μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου αρχικά. Άρα δεν μπορείτε να παρακολουθείτε απλώς το γεγονός ότι ένα σχέδιο πριν καν αρχίσει έχει δημιουργήσει προβλήματα. Υπάρχει θέμα κακοδιαχείρισης εδώ. Υπάρχει και κάτι άλλο από τις συζητήσεις. Θέλετε άμεσα αποτελέσματα δηλαδή προσανατολίζεστε στα αποτελέσματα. Ξέρετε ότι το ίτερ θα αποδώσει σε 50 χρόνια. Και τότε, εγώ θα έχω συνταξιοδοτηθεί όπως και εσείς, εκτός αν έχετε κάποια μαγική συνταγή. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο είναι σκόπο να ε, παγώσουμε αυτό το θέμα για τα επόμενα 10 χρόνια. Θα ήθελα τις απόψεις σας. Ωραία. Ε, αυτά για αυτό τον ε, γύρο. Ε, κυρία Καβάλιο. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να χαιρετήσω την παρουσία της Επιτρόπου και να τη συγχαρώ καθώς και τις υπηρεσίες της για το πολύ καλό έγγραφο σχετικά με τις πρωτοβουλίες, ε, τις καινοτόμες πρωτοβουλίες διότι εγώ χαιρετίζω ιδίως την κοινωνική πτυχή ε, και αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ε, ιδέα που δεν υπήρχε στα προηγούμενα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδίως όσον αφορά το δημόσιο τομέα και την καινοτομία στις δημόσιες υπηρεσίες. Η αδυναμία του εγγράφου αυτού αναφέρεται στα εργαλεία, τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να εφαρμοστούν αυτές οι αρχές. Και με ανησυχεί ιδιαιτέρως το θέμα των οικονομικών, χρηματοοικονομικών εργαλείων. Δεν έχουμε ευελιξία, έχουμε ε, προβλήματα με το ΙΤΕΡ και περιμένουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση του προϋπολογισμού διότι το έγγραφο το οποίο δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα είναι πολύ καλό έγγραφο αλλά αναφέρεται στον επόμενο προϋπολογισμό όχι στον τρέχοντα άρα προς το παρόν έχετε τον τρέχοντα προϋπολογισμό στο 2013 έχουμε λοιπόν ένα προϋπολογισμό ο οποίος είχε είχε καταρτιστεί προετών όταν θέματα σαν την καινοτομία ή το τι υφίσταται διαθέσιμο δεν ε, ε, ήταν αμφισβητήσιμο όπως και άλλα άλλωστε οι κλιματολογικές αλλαγές και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν αυτές τις πολύ σημαντικές προτεραιότητες για την Ευρώπη και αν αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις χωρίς να έχουμε κατάλληλα οικονομικά ε, μέσα μέχρι το 2013 ή το 2020. Γενικώ λοιπόν η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 θα μπορούσε να, να ε, χρηματοδοτηθεί σωστά το 2014. Έχετε προβλέψει κάποια λύση για αυτό το πρόβλημα. Αυτή είναι ουσιαστικά η ερώτηση την οποία ήθελα να σας απευθύνω. Ευχαριστώ. Έχω ακόμη δέκα ομιλητές που ζητούν το λόγο. Θα ήθελα όλους να σας παρακαλέσω να είσαστε πιο συγκεκριμένοι. Ο κύριος Βανίστρο είναι πρώτος. Ευχαριστώ. Σε αυτή τη φάση δεν νομίζω πως μπορούμε να βαθύνουμε. Νομίζω πως ο χαρακτήρας προσέγγισης που έχουμε τώρα είναι ολοκληρωμένος. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλά χαρτοφυλάκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι θετικό γιατί παίζεται ένα συντονιστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι η σύνδεση των εξωτερικών εταίρων σε αυτές τις εταιρικές ε, σχέσεις και το τι θα έπρεπε να γίνεται στα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί νομίζω ο καθένας να είναι στην πρώτη σειρά εάν δεν ε, ε, έχει και κάτι να προσφέρει. Κάτι το οποίο βεβαίω ήταν το πρόβλημα στην πολιτική της Λισαβόνας. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και πλέον αυτά τα μέσα τώρα για την χρηματοδότηση το έθεσαν και άλλοι το ερώτημα, αλλά βλέπω εδώ πέρα στα κείμενα της ε, ενδιάμεσης ε, αναθεώρησης πως μιλάμε για μια συνέργεια μεταξύ των διαφόρων κονδυλίων, κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Δεύτερον, κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον, η καινοτομία τώρα την οποία προτείνεται όσον αφορά την προσέγγιση του Κοινοβουλίου γιατί κάθε χρόνο ακούμε πως θα υπάρχουν αυτές ε, ή μεγάλες πρωτοβουλίες με εξωτερικούς εταίρους. Γιατί θα πρέπει να φροντίσουμε αυτός ο νέος διάλογος κάθε φορά που μας βγούμε στο πέρα στο Κοινοβούλιο και μιλάμε να μην είναι μόνο κάτι το οποίο υπάρχει στα χαρτιά αλλά να έχει ένα πραγματικό αντίκρισμα. Ευχαριστώ κυρία Χέρτσοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που ήρθατε και είστε σαφείς, μόνο οι γυναίκες το μπορούν αυτό. Οπότε συγχαρητήρια. Έχω να πω πολλά πράγματα, όχι πάρα πολλά, αν φοβάστε. Ένα από αυτά είναι ο προπολογισμό. Πώς μπορείτε να φέρετε το Συμβούλιο με το μέρος σας. Είδαμε τι έγινε με, το με τον προπολογισμό του 2011 και το κεφάλαιο έρευνας και ανάπτυξης, ε, ένα α συν, συν 5. Οπότε πώς μπορεί να μετακινηθεί το Συμβούλιο, γιατί χωρίς βεβαίως χρηματοδοτικά μέσα δεν θα επιτύχετε ούτε εμείς τους ε, στόχους μας. Μέχρι το 2014 θα έχει λήξει η δική μας η θητεία, η δική σας θητεία και θα πρέπει να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Γιατί δεν θα σταματήσει ο κόσμος επειδή διστάζει η Ευρώπη, οπότε είναι ξεκάθαρο πως πρέπει να προχωρήσουμε. Επίσης εγώ θα προτιμούσα να διαφωνώ με τους συναδέλφους για το ΙΤΕΡ. Συμφωνώ με αυτά τα οποία λένε. Αλλά αυτό ισχύει για οτιδήποτε είναι μεγάλο. Γαλιλαίο, GMS, ε, σχέδιο όλα αυτά. Οτιδήποτε είναι μεγαλύτερο από ένα κράτος μέλος και μικρότερο από 27 είναι πρόβλημα. Και το ΙΤΕΡ είναι ένα από αυτά τα έργα. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε παραδείγματος χάρη το καταλογό S-Free. Κατόπιν, επειδή είμαι Ουγγαρέζα. Ποια θεωρείτε ότι μπορεί να είναι μια πιθανή επιτυχία της ε, Ουγγρικής Προεδρίας όσον αφορά την Ένωση της Καινοτομίας. Ποια είναι τα σχέδιά για τους επόμενους 6 μήνες και η άποψη για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας που βρίσκεται στην Ουγγαρία. Θέλω να μάθω πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα για να έχει ως δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Πώς τα βλέπετε αυτά. Και σα ευχαριστώ που ήρθατε και εμεί θα σας βοηθήσουμε ω Κοινοβούλιο, ειδικά στη διαδικασία της συνδιαλλαγή. για να αποκαταστήσουμε αυτή τη γραμμή που έκοψαν για την έρευνα. Ευχαριστώ, Τόμψεν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, για την παρουσίασή σας κυρία Επίτροπε. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα, την ακούσαμε και φαίνεται ότι θα έχουμε έναν εξυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος. Το, κάτι το οποίο είχαμε αποπειραθεί αρκετό, από, καιρό, από αρκετό καιρό πριν μιλήσαμε για την καινοτομία για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες διασυνοριακά, διότι νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Έχει οριμάσει το πλαίσιο και θα πρέπει να μεταφέρουμε τις γνώσεις μας από τη μία χώρα στην άλλη χρησιμοποιώντας και τις πολιτισμικές μας αποκλίσεις και διαφορές. Ως προς τις δημόσιες προμήθειες και την καινοτομία υπάρχει μία χώρα από τις 27 όπου υπάρχει μία νομοθεσία για, την, για τις δημόσιες προμήθειες και την καινοτομία. Από όσο γνωρίζω, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2007, στο Υπουργείο Εμπορίου. Έχουν λοιπόν μεγάλη πείρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο υπόλοιπο της Ευρώπης. Μιλήσατε για ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Συμβουλίου, κάτι το οποίο με βρίσκει σύμφωνη. Θεωρείτε ότι το ε, Ευρωπαϊκό αυτό ερευνητικό συμβούλιο, συμβούλιο έρευνας θα πρέπει να έχει υψηλότερο προϋπολογισμό. Επίσης μιλήσατε για συνέργεια με το πρόγραμμα πλαίσιο. Θα πρέπει να υπάρχει συνέργεια των διαφόρων προγραμμάτων υποστήριξης, αλλά δεν είδαμε πολλά παραδείγματα. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να γίνει μία αξιολόγηση της συνέργειας μεταξύ των προγραμμάτων πλαισίων και των διαρθρωτικών ταμείων και αν υπάρχουν ε, δυσκολίες για να δημιουργήσουμε μία πλαισίωση. Εγώ είμαι συντονίστρια στην Επιτροπή Γυναικών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο θα δώσετε προτεραιότητα σε γυναίκες ερευνήτριες και αυτή τη στιγμή εκπονούμε μία έκθεση για την ισότητα των δύο φύλων στον τομέα της έρευνας. Η κυρία Χόλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επίτροπο για την λεπτομερή της ε, παρουσίαση για την Ένωση της Γενοτομίας. Τρεις ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Πρώτα απ' όλα, μετά από αυτά τα οποία είπε η κυρία Βίκη Φόρτ, γνωρίζουμε όλοι τις οικονομικές δυσκολίες ε, των κρατών μελών αυτή τη στιγμή. Πώς νομίζετε πως θα μπορέσει η Ένωση της Καινοτομίας και εν ευθέτω χρόνο το πρόγραμμα πλαίσιο 8 να βοηθήσει τη στιγμή που πάρα πολλές ε, πρωτοβουλίες αλλά επικαλύπτονται στα μελη Μπορείτε να μας πείτε πώς τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να γίνουν πιο αποτελεσματικά και να εστιάσουν τους περιορισμένους πόρους τους. Δεύτερον, η Ένωση της Κοινοτομίας αναφέρει το στρατηγικό σχέδιο ενεργειακής τεχνολογίας ως μία οριζόντια προσέγγιση σε μία αλλαγή για την κοινωνία. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο πώς το σχέδιο αυτό κολλάει με την ε, Ένωση της ε, Καινοτομίας. Θα ήθελα να το διευκρινίσετε αυτό. Και τρίτον, επίσης για το θέμα της, ε, των κοινωνικών αλλαγών, ένας από τους τομείς που αναγνωρίζετε πως είναι πάρα πολύ σημαντικός είναι η υγεία στην τρίτη ηλικία και αναρωτιέμαι πώς η ένωση αυτή της καινοτομίας θα βοηθήσει και εδώ πέρα μιλάω βεβαίως για την οδηγία κλινικών πειραμάτων. Νομίζω πως υπάρχει μια εξολόγηση αντικτύπων που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στην ε, Κομισιόν και αναρωτιέμαι εάν ε, ξέρετε ποιες είναι οι αλλαγές κλειδιά που θα προέκυπταν από μια τέτοια οδηγία. Τέλος, θα ήθελα βεβαίω να σας ευχαριστήσω γιατί αντιλαμβάνομαι πως το γραφείο σας ε, ασχολείται με ένα σχέδιο συνεργασίας για τα κλινικά πειράματα και σας ευχαριστώ για αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ε, παρουσίαση. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν μιλάμε για την πολιτική καινοτομία, νομίζω πως θα πρέπει να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί είναι ο κινητήρας ε, της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ μιλάμε για τα κονδύλια που πηγαίνουν στην έρευνα. Ελπίζω μαζί να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για το Γαλιλαίο. Δυστυχώς τα υπάρχοντα κονδύλια για δορυφορικά συστήματα πλοήγησης ε, δεν ε, θα μπορέσουμε να τα εκμεταλλευτούμε πλήρως, δηλαδή αναφέρομαι στο Γαλιλαίο, όταν ε, ολοκληρωθεί, εκτός εάν ε, δώσουμε τώρα τα απαραίτητα κονδύλια. Τώρα θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Θεωρώ πως ε, η συζήτηση θα ήταν ευρύτερη αν θα μπορούσατε να απαντήσετε το ερώτημα μου. Ξέρω πως ο χρόνος δεν επαρκεί. Το ερώτημά μου έχει να κάνει το εξής. Την τελευταία δεκαετία, δυστυχώς, η αποβιομηχάνηση ήταν αυτό το οποίο έλαμβανε χώρα στην Ευρώπη. Δηλαδή είχε τις εγκαταστάσεις καινοτομία ε, στην επικρατεία της Ένωση, αλλά η παραγωγή πήγαινε σε τρίτες χώρες ε, όπου ήταν μικρότερο το κόστος παραγωγής. Και τώρα υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή αποσυνδεθεί η καινοτομία από την παραγωγή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χάσει και την δυνατότητα καινοτομίας. Και το ερώτημα μου είναι το εξής. Πώς θεωρείτε πως θα πρέπει να συνδεθεί η πολιτική καινοτομίας με την βιομηχανική πολιτική της Ένωσης, γιατί εγώ πιστεύω πως συνδέονται. Και Εάν το μεγαλύτερο κομμάτι της ε, βιομηχανίας ε, πάει σε άλλες ε, περιοχές του πλανήτη, κινδυνεύει και η καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι θα μπορέσει να φύγει από την κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να σκεφτεί μια φιλόδοξη βιομηχανική πολιτική που θα είναι και οικολογικά αποτελεσματική για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε και καλές δουλειές στην Ευρώπη. Γιώργα Σίσελη. Έχετε τον λόγο. Όχι. Ο κύριος Όντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ακούτε τους βουλευτές και όλα τα προβλήματα τα οποία υποβάλλουμε. Τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα για το ίτερ. Θα ήθελα να σας πω πως υπάρχουν δύο πράγματα για τα οποία θλίβομαι. Πρώτα απ' όλα το ότι οι πτυχές ε, του προϋπολογισμού φαίνονται πως είναι αυτό το οποίο μετράει και δίνει τον τόνο ε, σε αντίθεση με την πτυχή της ε, τεχνολογίας. Θα ήθελα να πω λοιπόν πως δεν θέλουμε η Επιτροπή Προϋπολογισμού να δώσει εδώ πέρα τον τόνο. Εμείς ως ευρωβουλευτές βεβαίως ασχολούμαστε με το Ίντερ. Θα ήθελα, όπως σας είπα, να προβώ σε δύο υποδείξεις. Ξέρουμε ότι βρίσκουμε πάντα την λύση των ζητημάτων στην επιστήμη όταν μιλάμε για θέματα καινοτομία, διότι ε, δεν μπορούμε παρά να είμαστε δεοντολόγοι όταν μιλάμε για θέματα επιστημών και έρευνα, έρευνας. Θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το ηθικό μήνυμα, το ηθικό δίδαγμα, όπως τονίσατε και εσείς. Η συνάδελφος Χολ μας μίλησε για κοινοτικοποίηση της πολιτικής έρευνας που είναι ένα στοιχείο ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς σε διαπραγμάτευση με τα κράτη-μέλη για να δούμε πώς στην Ήπειρο ως προς την ε, Τελωνιακή Ένωση, την άμυνα, τις στρατιωτικές δυνάμεις και την έρευνα μπορούμε να φτάσουμε σε ένα κοινό παρονομαστή. Θα πρέπει να γίνει μία έρευνα, ένας απολογισμός των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να προβούμε σε έναν ισολογισμό που θα αναλάβει το ελεγκτικό συνέδριο και τα 27 εθνικά ελεγκτικά συνέδρια για να δούμε πώς μπορούμε να κοινοτικοποιήσουμε την ερευνητική πολιτική και να ε, προβούμε σε εξοικονόμηση τη στιγμή που το δημόσιο χρήμα σπανίζει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, δέχομαι πολύ θετικά την παρέμβασή σας διότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τον τομέα της καινοτομία της έρευνας, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, για να ανταποκριθούμε σε συνεκτικές πολιτικές ως προς το περιβάλλον. Τώρα, ως προς το πρώτο ερώτημα στην Ένωση για την Καινοτομία προβλέπεται αύξηση των δημοσίων και ιδιωτικών δαπανών και νέα μέτρα για την καλύτερη προσπελασιμότητα, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ. Τι θα γίνει με αυτές που θέλουν να επενδύσουν στον τομέα της έρευνας. Ως προς τα διαρθρωτικά ταμεία, έχει μεγάλη σημασία η συνέργεια των επιμέρους προγραμμάτων. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την ε, χρήση αυτών των πόρων. Τέλος, τρίτο ερώτημα. Οι εθνικές πολιτικές γνωρίζουν δραστικές περικοπές στον τομέα της έρευνας, μιλώντας για ένα μεγάλο έλλειμμα στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει μεγάλη αποδυνάμωση. Όμως γίνεται λόγος για 3,7 εκατομμύρια θέσεων εργασίας μέχρι το 2020. Πώς τόσο αποκλίνουσες πολιτικές μπορούν να πραγματοθούν αν λάβουμε υπόψη και την εκπαιδευτική πολιτική των κρατών μελών. Πώς μπορούν να συγκλίνουν η εκπαίδευση και η έρευνα. Και εδώ αναφέρομαι ιδιαίτερα στους νέους ερευνητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την ε, Επίτροπο. Θα ήθελα να εκφράσω μία σκέψη και μία ε, ερώτηση. Σήμερα είδα μία διαφήμιση στο αεροδρόμιο και μιλούσε για το τελευταίο χάμπουργκερ Jack Daniels. Το απόλυτο, ναι. Ξέρω τι σημαίνει hamburger, αλλά όταν μιλάμε για το the ultimate Jack Daniels hamburger, τι εννοούμε. Ζούμε σε ε, μία εποχή όπου δεσπόζει η υπερβολή. Υπάρχει όμως ένας στόχος, τον οποίο ακόμα δεν έχουμε φτάσει, δηλαδή το στόχο της ε, συνθήκης της Λισαβόνας να έχουμε την πλέον ανταγωνιστική οικονομία. Τώρα μιλάμε ε, για, την, για το τομέα της ανταγωνιστικότητας. Ε, και εδώ ισχύει η διαφήμιση το The Ultimate Jack Daniels Hamburger. Και εδώ υπάρχει ένα στοιχείο υπερβολής δεν μπόρεσα να επεξηγήσω καμία ευρωπαϊκή στρατηγική σε κανέναν ψηφοφόρο. Ποτέ, μα ποτέ. Άρα μιλάμε για μεγαλόπνοα και μεγαλόστομα σχέδια τα οποία δεν οδηγούν πουθενά. Δεν υποτιμούμε όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν ένα, μια εγγενή δυναμικότητα. Τη στιγμή που μιλάμε για λιτότητα για τις ε, εθνικές κυβερνήσεις που θα έχει επιπτώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι νόημα έχει και πώς μπορεί να ε, προωθηθεί πραγμάτωση αυτών των στόχων. Η συνάδελφος Τόγια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επίτροπο για αυτή την εισήγηση γιατί καταβάλετε μια μεγάλη προσπάθεια να δούμε και την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Μας ενδιαφέρουν νέα απλουστευμένα ε, σχέδια και μέθοδοι, γιατί πολλές φορές οι στόχοι μας είναι θετικοί, αλλά απέχουμε πόρο από τα κατάλληλα μέσα και μας ενδιαφέρει και η αποτελεσματικότητα των ε, μέσων και μέτρων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε αυτούς τους δείκτες και θα δω τι ε, απάντηση θα δοθεί στο θέμα των ε, δικτών. Στο ερώτημα που υπέβαλε μία συνάδελφος. Νομίζω λοιπόν ότι η προσέγγιση είναι πολύ θετική επειδή μιλάμε για μεθοδολογία και προτεραιότητα επιλογών και επειδή καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια να επικεντρωθούμε στις μεγάλες προτεραιότητες, θα πρέπει να έχουμε συγκέντρωση δυνάμεων. Αυτό αφορά συνέργεια κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για, τα joint, για το joint programming και δεν ξέρω κατά πόσο εδώ θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, διότι μιλάμε για μεγάλες έρευνες στον τομέα της υγείας και υγιεινής και νομίζω ότι μόνο με μία συγκλίνουσα συνδρομή των κρατών μελών μπορούμε να προβάλλουμε την καινοτομία και την έρευνα, επί του πρακτέου δηλαδή διότι πολλές φορές βλέπουμε ότι μένουμε πολύ πίσω ως προς την έρευνα σε σχέση με άλλες ε, περιοχές του κόσμου. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε στις ΗΠΑ. Εάν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση προβεί στη σύσταση δικών της σχεδίων, θα είναι πιο ευέλικτη. Εάν απλώς συντονίζει τα, συντονίσει τα προγράμματα στα πλαίσια του joint programming, δεν θα καταφέρουμε και πολλά. Και δεύτερον, όπως είπε ο συνάδελφος μιλώντας για θέματα ηθικής δεοντολογίας, καινοτομίας και έρευνας, θα πρέπει να δούμε και την κοινωνική πτυχή του ζητήματος. Θα πρέπει να μας απασχολήσει η κοινωνική καινοτομία έτσι ώστε να πειραματιστούμε για τα νέα μοντέλα παραγωγής, γιατί υπάρχουν και νέα επαγγέλματα τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κοινωνική μας ζωή. Άρα η κοινωνική καινοτομία είναι ύψης της σημασίας και θα πρέπει να μας απασχολήσει περαιτέρω. Τελευταίος κύριος Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την εισήγησή της ως προς αυτό το έγγραφο. Θα ήθελα να δείξω ένα πρόβλημα που αφορά τις υποδομές στην έρευνα. Συμφωνώ απόλυτα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, διότι φαίνεται ότι είμαστε ουραγοί των ΙΠΑ και της Ιαπωνίας σε σχέση με τις επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας. Και αυτό θα μπορούσε να θέσει ένα πρόβλημα στο μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μόνος τρόπος να ανακτήσουμε δυνάμεις και να βραχύνουμε τις αποστάσεις με τις ΙΠΑ είναι να προωθήσουμε την έρευνα σε όλα τα κράτη-μέλη για να προωθήσουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, να ασχοληθούμε και με την εξειδίκευση και την διαφοροποίηση στον τομέα της εξειδίκευσης. Δυστυχώς, τα νέα κράτη-μέλη δεν έχουν τις ε, κατάλληλες υποδομές. Και θα ήθελα να ρωτήσω την Επίτροπο κατά πόσο προβλέπει μία στρατηγική που να συνδυάζεται με την στρατηγική 2020 σε σχέση με την ε, ενίσχυση των υποδομών ερεύνης στα νέα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να έχουμε την καλύτερη δυνατή υποδομή και στα νέα για να υπάρχει ισομέρεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχω ακόμη μία δεύτερη ερώτηση του συναδε... της συναδέλφου Ναι, ε, ευχαριστώ. Ξέχασα τα μαγικά λόγια και συνεχίζει αγγλικά. Προτού τελειώσω με αυτό η κυρία Μέρκες. Κυρία Επίτροπε, έχετε συνεργαστεί πολύ στενά με τον Επίτροπο Ταγιάννη και αυτό είναι πολύ καλό διότι κατά αυτόν τον τρόπο συνδυάζεται την έρευνα με τις επιχειρήσεις. Ε, πρόκειται κάποια στιγμή να μας πει ε, τη δικιά του άποψη από την άλλη πλευρά του φράχτη για το πώς και αυτός θα καλύψει και θα προωθήσει την καινοτομία γιατί καλό θα ήταν να δούμε και τις δύο πτυχές. Και επίσης αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό κυρία ε, Επίτροπε σας ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια και εγώ προσβλέπω στη συνεργασία μας. Είναι μια πολύ βασική ε, στρατηγική, δεν ε, πρόκειται για πρόθεση των ε, και του Μακδόναλτ, ούτως ή άλλως εγώ είμαι φυτοφάγος. Αλλά ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις και προσβλέπω στη συνεργασία μας. Ωραία. Τώρα έχει το λόγο η κυρία Επίτροπος, εφόσον έχει ακούσει τις διάφορες ερωτήσεις και πρέπει να βρει κάποιο τρόπο εν το του δυνατού να τις απαντήσει εκτός και αν πρόκειται να ξανασυζητήσουμε για το ίδιο θέμα στην επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν όντως πολύ ενδιαφέρον για μένα και μου θύμισε τη συζήτηση που είχαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ομάδα καινοτομία στην Επιτροπή όπου προείδρευα όταν καταρτίζαμε την ανακοίνωση. Υπήρχαν αντικρουόμενες απαιτήσει, ανταγωνιστικές απαιτήσει και στο τέλος χρειάστηκε να συνοψίσουμε όλη τη συζήτηση σε ένα έγγραφο το οποίο είχε ξεκινήσει ε, και έπρεπε να είναι φιλικό προς το χρήστη για να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε αλλά συγχρόνως να είναι ουσιαστικό. Όλα αυτά λοιπόν αντικατοπτρίζουν επακριβώς ότι έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από, το, την Άνοιξη. Ε, βέβαια έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με τον Αντώνιο Ταγιάννη και απαντώ ξεκινώ από την τελευταία ερώτηση, ο οποίος τώρα καταρτίζει την δικιά του ανακοίνωση ε, για την βιομηχανική καινοτομία. Flagship σαν ε, ναυαρχίδες θεωρούνται και οι δύο αυτές ανακοινώσεις και θα ε, παρουσιάσει τη δικιά του ιδέα. Για να ξεκινήσω με το πιο δύσκολο θέμα από όλα τα οποία χρειάστηκε να αντιμετωπίσω από όταν έγινα επίτροπος είναι το θέμα του Twitter. Τώρα οι, τα ορυκτά καύσιμα καλύπτουν τα 80% των αναγκών μας, άρα συμβάλλουν στις κλιματολογικές αλλαγές ε, ως πλήστων και καλύπτουν και 80% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το Συμβούλιο συμφώνησε το 2009 ότι έπρεπε ε, να μειώσουμε τις εκπομπές από 80% 95% μέχρι το 2050 που είναι μια τεράστια πρόκληση για όλους μας διότι όλοι πρέπει να εμπλακούν σε αυτή την πρόκληση και είναι ε, μια πρόκληση και για το μέλλον της Ευρώπης και όπως σας είπα το είπα και στην ακρόασή μου αλλά δεν υπάρχει μη χρυσή λύση για να βρούμε την βέλτιστη μέση οδό για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε όλες ε, τις θετικές προοπτικές οι οποίες διαγράφονται. Δεν νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να διαγράψουμε την, ε, ε, την ενέργεια από καύσιμα για αυτόν τον τρόπο. Πολλά εξαρτώνται από το και όπως είπε και η κυρία Ντελκαστίγιο είναι ένα τεράστιο εγχείρημα και είναι φυσικό και αναμενόμενο ότι ένα πρόγραμμα τόσο περίπλοκο όσο το ΙΤΕΡ ε, συνεπιφέρει και ε, κινδύνους αλλά και προκλήσεις και από το Φεβρουάριο προσπαθούμε να θέσουμε το ΙΤΕΡ επί μίας ορθής και υγιούς βάσεως και οι δυσκολίες δεν έχουν μόνο σχέση με τις χρηματικές δυσκολίες υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα προβλήματα για την διακυβέρνηση του ΙΤΕΡ και του ΕΦΟΡΙ ε ε. και εις ε, τη Βαρκελόνη είπαμε ότι συμφωνήσαμε να επιλύσουμε τα θέματα της διακυβέρνησης. Την πρώτη φορά που πήγα το Μάρτιο ή τον Απρίλιο στις Ηνωμένε Πολιτείε, το ίτερ ήταν ένα θέμα το οποίο ε, συζήτησα με τον ε, Υπουργό κύριο Ντιού διότι ε, το θέμα α, της δεσμεύσεώς μας για το ίτερ παραμένει το ίδιο αλλά για να προχωρήσει πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά να καταρτήσουμε τη σωστή διακυβέρνηση και έγιναν αλλαγές και στο Συμβούλιο του Ίτερ και στο ΕΦΟΑΡΗ. Αλλά ε, το Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε αλλαγές, να βρει λύσεις στα πλαίσια του, ε, των περιορισμών και μέσα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Έπρεπε δηλαδή όλη η χρηματοδότηση να γίνει από το το πρόγραμμα πλαίσιο 7. Πράγμα το οποίο για μένα δεν ήταν ε, δυνατόν. Δηλαδή το, ε, το πρόγραμμα πλαίσιο 7 δεν μπορούσε ε, να πιεστεί στο σημείο για να καλύψει όλες αυτές τις ε, ανεπάρκειες και γι' αυτό τις ελλείψεις. Και θεωρήσαμε ότι η πρόταση που διατυπώσαμε ήταν ισοσκελισμένη, δίκαια και θέλουμε η πρόταση αυτή να εφαρμοστεί. Θα ήθελα λοιπόν να με στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προωθήσουμε την πρόταση αυτή. Διότι όπως είπα θεωρώ ότι είναι και δίκαιη και ισοσκελισμένη και είναι η μόνη η οποία θα μπορέσει να προστατεύσει τις κοινέ μας προτεραιότητες είναι μία συζήτηση η οποία συνεχίζεται στα διάφορα θεσμικά όργανα, μπορεί να, να συνεχιστεί και επί αρκετό καιρό. Αλλά πρέπει ε, να σεβαστούμε ότι οι δύο πλευρές των νομοθετικών οργάνων θα βρουν κάποια λύση ε, η οποία θα μπορέσει να εξελιχθεί περαιτέρω. Αυτό που πρέπει επίσης να πω, ένα πράγμα το οποίο Λοιπόν ζητήσαμε και εσείς μου ζητήσατε συγκεκριμένα είναι να μπορέσουμε να περιορίσουμε το κόστος στο FOE και ε, για να αναπτύξουμε ορισμένα μέρη από αυτό το τεράστιο πρόγραμμα ήδη έχουμε εξοικονομήσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι σημαντικό διότι το κοστολόγιο σε σχέση με ε, τα ε, τμήματα ε, και τα ανταλλακτικά τα οποία ζητούσαν έχει μειωθεί και άρα το ο κόστος για το ίτερ και για το ΕΦΑΗ e έχει μειωθεί επίσης. Αν θέλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε την δημιουργία του θα χρειαστούν ε, μεγάλες ε, μεταφορές από τα εργαστήρια, από τα ε, εργοτάξια στα εργαστήρια και θα πρέπει να υπάρξει μία περιστολή που είναι πολύ σημαντική διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και τα κράτη-μέλη αμφισβητούν πάρα πολύ στη θέση της απασχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν ε, να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε και τη δυνατότητα ανακαίνησης αλλά και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Χωρίς λοιπόν να θέλω να αναφέρομαι σε κάθε ευρωβουλευτή ονομαστικά, θα απαντήσω συνολικά πολλές φορές σε διάφορες ερωτήσεις μαζί. Καταρχήν όσον αφορά τις συνεργασίες. Ο στόχος των συνεργασιών είναι διτός. Αφενός να συνδυάσουμε τους πόρους και τις δυνάμεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κρατών μελών, βιομηχανίας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα ιδίως στους τομείς που ενδιαφέρουν το κοινό. Και οι προκλήσεις αυτές δεν είναι απλώς μόνο προκλήσεις αλλά και θαυμάσιες ευκαιρίες ε, για ε, νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικές και για δυνατότητες που ανοίγονται και μπορούν να προσφερθούν στην παγκόσμιο αγορά. Ε, βέβαια η βάση της Ευρώπης πρέπει να είναι βιομηχανική, να δημιουργήσει δημιουργήσει νέες αηφόρες θέσεις εργασίας σε ένα πρόσφορο μέλλον. Και ε, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Ουσιαστικά για να λύσουμε δύο προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή μας εμποδίζουν. Το πρώτο είναι το θέμα το οποίο ετέχθη από όλους τους ομιλητές σχεδόν ότι υπάρχει υπερβολικός κατακαιρματισμός. Δηλαδή τα διάφορα εργαλεία και σε επίπεδο ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κράτους μέλους πολλές φορές ε, ε, δεν συνεργάζονται αντί να ενισχύουν το ένα στο άλλο και ε, έτσι χάνουμε πολύτιμες ευκαιρίες. Για να λύσουμε λοιπόν αυτό το κατακαιρματισμό των συνεργασιών θα απλοποιήσουμε καλύτερα και θα ενισχύσουμε τις διάφορες δυνατότητες τα κοινά προγράμματα, τις ηγετικέ αγορές ε, και τις πλατφόρμες ε, όπως και τα ταμεία. Επίσης δεν φτάνει να ε, οδηγηθούν αυτές οι καινοτομίες στην αγορά. Η ιδέα από τις συνεργασίες είναι να καταργήσουμε τα εμπόδια στο σύστημα συνεργασιών και καινοτομίας, δηλαδή τα θέματα της

Ε, αποδοχής ε, της ε, τυποποίησεως όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν τις δημόσιες προμήθειες διότι υπάρχουν, υπάρχουν πολλές σωστές ιδέες οι οποίες όμως δεν φτάνουν στην αγορά για να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις γιατί να μην ξαναδούμε αυτές τις δυνατότητες συνδυάζοντας με την έρευνα η οποία θα συνεχίζεται για να κερδίσουμε χρόνο και αφετέρου άπαξ και υπάρξει η πρόοδος το κοινό να μπορέσει να υποφεληθεί το ταχύτερο δυνατόν. Και η μαγική λέξη είναι ταχύτητα, διότι οι αρχηγοί κρατών ε, το συζητήσουν όπως ξέρετε το Δεκέμβριο και το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητος είχε μια εξαιρετική πρώτη συζήτηση στην τελευταία μας συνεδρίαση και τα συμπεράσματά του θα ε, διατυπωθούν τέλη Νοεμβρίου στο επόμενο Συμβούλιο Ανταγωνιστικό. Είμαστε υπέρ της ιδέας της συνεργασίας και αυτή τη συνεργασία την οποία προσπαθούμε να προωθήσουμε στη δραστήρια και αποδοτική γύρανση. Δηλαδή να υπάρχει ο στόχος να έχει κανείς δύο επιπρόσθετα χρόνια πρόσφορα και υγιή μέχρι το 2020. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι μπορούν να κατανοήσουν και να αποδεχθούν οι πολίτες και θα υπάρχουν πακέτα εργασίας τα οποία θα πρέπει να συνδυαστούν. Δηλαδή να ευρεθούν και να αναπτυχθούν καινοτόμες ε, ενέργειες, φάρμακα και θεραπείες για ε, να καταπολεμήσουν τις ασθένειες που συνδυάζονται με την γύρανση ή ε, να υπάρξουν βιώσιμες λύσεις για την παρακολούθηση των ηλικιωμένων διότι πολλές φορές λέγεται ότι η υγιής γύρανση είναι, δεν είναι πραγματικά συνεργασία εγώ διαφωνώ διότι μπορείτε να πείτε ότι είναι κάτι μαλακό και ε, όχι πολύ απτό αλλά υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για τις εταιρείε σε αυτό το τομέα και ήδη στην γεωργία και στο ICT ε, έχουμε πολλές τέτοιες δυνατότητες διότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας ε, για να υπάρχουν οι πρωτοβουλίες ε, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν ανεξάρτητες ζωές με καλύτερη υγεία και είναι πολύ βασικό αυτό το θέμα διότι αποδυναμώνει τα δημόσια οικονομικά και εμείς θέλουμε να βελτιωθούμε βελτιωθεί η κατάσταση γιατί όλοι γερνάμε, θέλουμε να γερνάμε πιο υγιώς, να ζούμε ανεξάρτητα και να υποφεληθούμε από αυτές τις δυνατότητες. Η οικονομική λοιπόν λογική για αυτή τη συνεργασία είναι ε, πολύ θετική, θα συνδράμει την βιομηχανία διότι υπάρχουν ε, νέες και αναπτυσσόμενες αγορές, οι άνθρωποι θα είναι πιο υγιείς, πιο παραγωγικοί για περισσότερο καιρό και για τα κράτη-μέλη το βασικό θέμα για αυτούς είναι να μειωθεί το κόστος περιθάλψεως των ασθενών που αποδυναμώνει τα δημόσια, τους δημόσιους προϋπολογισμούς. Ελπίζω λοιπόν ότι θα στηρίξετε και την ιδέα της συνεργασίας και την πιλωτική συνεργασία. Βέβαια υπάρχει μία νέα δυνατότητα μια νέα προσέγγιση, κάτι το οποίο δεν είχαμε κάνει. Γι' αυτό ήθελα μια πιλωτική συνεργασία για να μπορούμε να συνεργαστούμε στενά με όλους τους ενδιαφερόμενους, με το Κοινοβούλιο βεβαίως, στην πιλωτική αυτή φάση. Η πιλωτική φάση το επόμενο καλοκαίρι θα οδηγήσει σε μια ανακοίνωση, μια ανακοίνωση η οποία θα αντλήσει κάποια διδάγματα και θα ορίσει πώς θα λειτουργούν αυτές οι συνεργασίες στην πράξη. Μπορώ να πω ήδη όμως πως δεν μιλάμε για μία νέα υπηρεσία ή κάτι τέτοιο, αλλά μιλάμε για μία ευκίνητη πολιτική δομή για να κατευθύνει τις συνεργασίες, στην οποία θα εμπλέκεται πλήρως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε δεν μιλάμε για νέα υπηρεσία ή για κάτι καινούριο το οποίο θα καταστήσει ακόμη χειρότερο το γραφειοκρατικό άρθος. Τώρα, αν μπορεί να είναι πιο καινοτόμο ο δημόσιο τομέα. Εγώ πιστεύω πω οπωσδήποτε μπορεί. Υπάρχει ένα κλίμα, όπως ξέρετε, δημοσιονομικής ε, λιτότητας σε όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε ο δημοσιοτομέας πρέπει να μπορέσει να επιδείξει μεγαλύτερη καινοτομία για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσει ε, και προσδοκίες των χρηστών του δημόσιου τομέα. Οπότε, η Ένωση της Καινοτομίας ε, ζητά μια καλύτερη κατανόηση του τι είναι ο καινοτόμος δημόσιου τομέας και βεβαίως θα πρέπει να διαφημίσουμε περισσότερο επιτυχείς πρωτοβουλίες και την ε, μετρήσιμη πρόοδο. Είπα λοιπόν στην αρχή, κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου, πως η Κομισιόν ε, θα ξεκινήσει αυτή, ε, τον πίνακα βαθμολογίας καινοτομία του δημοσίου τομέα ως βάση συγκριτικής αξιολόγησης, αλλά πέρα από αυτό, από το επόμενο έτος, η Κομισιόν θα υποστηρίξει ένα πρόγραμμα έρευνας για το δημόσιο τομέα και την κοινωνική καινοτομία που θα δει ζητήματα όπως η παρακολούθηση, η αξιολόγηση, και πιθανά εμπόδια στην καινοτομία. Και επίσης σκοπεύουμε να εξερευνήσουμε με τα κράτη-μέλη την δυνατότητα δικτύωσης ηγετών του δημοσίου τομέα για να μπορέσουν αυτοί να ανταλλάξουν τις βαλιστές πρακτικές. Και νομίζω πως η Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή θέση για να μπορέσουν να καταφέρουν να έρθει σε επαφή, να έρθει σε επαφή η και να διαδοθεί αυτή ακριβώ η πληροφορία που αφορά την καινοτομία, κάτι το οποίο έχει ζωτική σημασία για τους υπαλληλού και διοικητέ εκείνους του δημοσίου τομέα που θα εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές. Επίση θεωρώ πω δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το δυναμικό που υπάρχει για την δημόσια προμήθεια καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών. Γιατί αυτό είναι νομίζω ένας τρόπος να έχουμε πιο αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες. Τώρα βεβαίως δεν υπάρχουν στόχοι για τις δημόσιες προμήθειες, αλλά νομίζω πως τα κίνητρα τα οποία θα ευνοήσουν τις λύσεις ε, που αναλαμβάνουν κίνδυνο συχνά έχουν μια έλλειψη κατάρτιση και συχνά οι δημόσιες προμηθείες δεν θεωρούνται ένα εργαλείο πολιτικής και αυτή είναι μια ευκαιρία να, τα... να χρησιμοποιήσουμε ω τέτοιο. Και βεβαίω το έγγραφο το σχετικό ζητά από τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να αφιερώσουν ε, κομμάτι του προπολογισμού του γι' αυτό. Οπότε θα βασιστούμε εδώ πέρα στην εμπειρία του κοινού προγραμματισμού, με βάση την εμπειρία που είχαμε στην ευρωεκφυλιστικές ασθένειες. Επίσης θα συνδεθεί καλύτερη ατζέντα της έρευνα με το κομμάτι της καινοτομίας, έτσι ώστε η επιστημονική πρόοδος να μεταφραστεί πιο γρήγορα στα προϊόντα και υπηρεσίες που χρειαζόμαστε. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πήγα σε ένα συνέδριο το οποίο με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Το συνέδριο της Ένωσης Ιταλικών Βιομηχανιών. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ακόμη μικρότερες κλίμακας, μικρές εταιρείες, με τρία ή πέντε άτομα που δουλεύουν ε, και θέλουν βεβαίω να καινοτομήσουν, αλλά δεν έχουν εργαλεία ή ένα σύστημα στήριξη για να κάνουν κάτι τέτοιο. Και εντυπωσιάστηκα από τον αριθμό μικρών εταιριών που έδωσαν πρακτικά παραδείγματα του που κάνουν εξαιρετικά πράγματα και τα οποία εξάγουν τελικά για να αναπτυχθούν σε άλλες χώρες. Και όπως όλοι ξέρουμε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και πολλά από τα μέτρα που ανακοινώσαμε στην, ε, στο έγγραφό μας ε, θα ωφελήσουν αυτές τις επιχειρήσεις. Αναμένουμε και άλλα μέτρα τα οποία θα ωφελήσουν τις μικρομισές επιχειρήσεις, όπως παραδείγματος χάνει τη βελτίωση πρόσβασης στην χρηματοδότηση της καινοτομίας, κατά το οποίο είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη και σε ολόκληρη την Ένωση. Και νομίζω πως αύριο θα έχετε την ευκαιρία, εάν θυμάμαι καλά, να συζητήσετε με την κυρία Έρικα Μάν και τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνα. να συζητήσετε το μέσο RSFF, το οποίο είναι μια εξαιρετική επιτυχία και προσπαθούμε να το επεκτείνουμε, να το αλλάξουμε για να συμπεριλάβει περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε οι γενικές αρχές και η πολιτική που ακολουθεί το ΑΣΦΕΦ νομίζω είναι εξαιρετικά επιτυχής και κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα κύριε Πρόεδρε είναι να απελευθερώσουμε την επόμενη δόση κονδυλίων ε, και θα δείτε αύριο γιατί ε, αυτό αυτή τη στιγμή είναι κατεπήγον βεβαίως άλλα μέτρα πρέπει να απλοποιήσουμε τα μελλοντικά προγράμματα έρευνας και χρηματοδότηση. αυτό θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διευρύνουμε το εύρος της ευρωπαϊκής πολιτικής καινοτομίας πέρα από την τεχνολογική καινοτομία και να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μη τεχνολογικούς τομείς. Και εδώ πέρα θα ήθελα να επαναλάβω το ε, σύσταση να του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Βιομηχανίας ε, και του πιλωτικού έργου κοινωνικής καινοτομία και εκεί πέρα βεβαίω θα βοηθήσουμε πάρα πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα υπάρχοντα σχέδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν πως η συνεισφορά του κοινοτικού προϋπολογισμού μπορεί να μοχλεύσει, αν θέλετε, ένα εικοσαπλάσιο κεφάλαιο από τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε θέλουμε ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει διασυνοριακά Κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου, θέλουμε να ενισχύσουμε την διασυνοριακή επαφή καινοτόμων εταιριών με επενδυτές γιατί τι σημαίνει έχουμε μια ε, καινοτόμο επιχείρηση εδώ και κάπου αλλού επενδυτή και δεν συναντιόνται ποτέ. Οπότε θα πρέπει αυτά τα δύο να συναντηθούν. Επίσης αξίζει να σημειώσουμε πως το Φόρουμ Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων θα αποτελέσει πλατφόρμα ανείχνευσης αυτών των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ειδικά οι μικρές και καινοτόμες επιχειρήσεις. Συνολικά λοιπόν υπάρχει έμφαση στο πώς θα αναμειχθούν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς θα τις βοηθήσουμε να γίνουν, να εμπλακούν ακόμη περισσότερο. Σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να πούμε πως οι μεγάλες συμφωνίες που υπογράφηκαν πριν από την 1η Οκτωβρίου δείχνουν πως 5.269 συμμετέχονται συμμετοχές μικρομεσαίων επιχειρήσεων από 4.100 διαφορετικούς ε, ε, δικαιούχους και είχαμε 1.459 Μικρομισέ επιχειρήσει που αποτελούν ένα 14% τη συνολικής χρηματοδότηση. Οπότε το ποσοστό το οποίο πηγαίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται σταθερά από την αρχή του προγράμματος πλαισίου 7. Για να δω τώρα. Διεθνή συνεργασία, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το συνεχίσουμε για την τυποποίηση και την διεθνή συνεργασία. Ένα από τα ζητήματα το οποίο, τα οποία έθιξα στην επίσκεψή μου στις ΗΠΑ ήταν πως εάν δεν θέσουμε παγκόσμιες προδιαγραφές στην Ευρώπη και στην Αμερική, αυτό θα γίνει στην Ανατολή, κάτι το οποίο δεν θα θέλαμε. Οπότε πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε στον ανταγωνισμό μεταξύ μας και να βρούμε τρόπους συνεργασίας για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω πως θα δείτε τους επόμενους μήνες μια επανεξέταση του πώ ορίζονται οι προδιαγραφέ και βεβαίω ο Επίτροπο ο κ. Σταγιάννη που είναι υπεύθυνο για αυτόν τον τομέα θα το προωθήσει αυτό με τρόπο στοχευμένο. Τώρα για το πώς θα μείνουν οι ερευνητές εδώ και πώς ε, θα αναπτύξουν δυνατότητες καριέρας και γενικότητας. Αυτό ήταν κάτι που πάντα μας απασχολούσε. Και την προηγούμενη επιτροπή, ο προκατοχός μου, ο κύριος Ποτότσνικ, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με αυτό το θέμα. Είναι κάτι που με ανησυχεί γιατί θεωρώ πως ε, Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα, αναφέρθηκε αυτό και με τις γυναίκες ερευνήτριες, υπάρχει λοιπόν μια διαρροή αν θέλετε. Πολλοί ξεκινάνε, με, πολλές γυναίκες ξεκινάνε, μετά σταματάνε να κάνουν οικογένεια και βεβαίως το περιβάλλον δεν επιτρέπει την ενσωμάτωσή τους αφού έχουν φύγει. Οπότε πρέπει να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για να μπορέσουν να επανέλθουν οι γυναίκες, αλλά πρέπει να διευκολυνθεί η ζωή του ερευνητή στην Ευρώπη να γίνει πιο φιλική προς την οικογένεια έτσι ώστε αυτοί οι υπέροχοι ερευνητές που έχουμε να θέλουν να ζήσουν και να δουλέψουν εδώ και να ενθαρρύνουμε και ερευνητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να έρθουν να δουλέψουν εδώ πέρα. Επίσης θεωρώ πως είναι θετικό να ταξιδεύουν, να πηγαίνουν στο εξωτερικό ερευνητέ, αλλά εγώ θα ήθελα να επιστρέφουν εδώ πέρα. Και θα ήθελα να υπάρχουν κάποια μέτρα ε, που να τους ενθαρρύνουν. Και βεβαίως όταν έχουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, όπως μας επιτρέπει τώρα η συνθήκη της Λισάβονας, θα έχουμε ένα πλαίσιο για τους ερευνητές για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τους καλύτερους και να τους κρατήσουμε εδώ πέρα, να δουλέψουμε εδώ. Για το RSFF το είπα απλοποίηση. Η έκθεση της κυρίας Καρβάλιο ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε στην απλοποίηση. Νομίζω πως τόνισε πολλά από τα στοιχεία της απλοποίησης που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχουμε ήδη τρεις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχουμε λάβει με την ανακοίνωση περί απλοποίησης, με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και βέβαια το ανεκτό ποσοστό σφάλματος. Ξέρω πως ειδικά ο κύριος Σοντή έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για το ανοιχτό, ανοιχτό κίνδυνο σφάλματος, γιατί δεν είναι κάτι το εύκολο. Ίσως είναι ε, εύκολο σε αυτή την επιτροπή, αλλά όχι τόσο εύκολο σε μία από τις αδελφές επιτροπές. Αλλά είναι ένα θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα είναι σημαντική η διαφορά εάν έχουμε τους ερευνητές και τους επιστήμονες να μην ασχολούνται με το να συμπληρώνουν έντυπα στα γραφεία τους και να μπορούν να είναι στα εργαστήρια για να κάνουν την πραγματική τους δουλειά. Επίσης, να διασφαλίσουμε πως οι ελεγκτές μας στη Γενική Διεύθυνση δεν ασχολούνται και τρώνε το χρόνο τους με το να εξετάζουν τα τελευταία μικροποσά για να πάει το νούμερο κάτω από το 2%. Θεωρώ λοιπόν πως το, ανεκτό, ο ανεκτός κίνδυνο ασφάλματος είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση και είναι κάτι ε, το οποίο μας απασχολεί και ξέρω πως και τα μέλη που είναι και στις δύο επιτροπές ε, εργάζονται λεπτομερώς για να καταλήξουμε σε μια λύση. Όμως παράλληλα πιστεύω και αυτό το εθιξαν έθιξαν ορισμένα κράτη-μέλη σε σχέση με το σχετικό κόστος, το εμπλεκόμενο κόστος. Προσπαθούμε να εξεύρουμε λύσεις έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα στο σύνολό του. Επίσης, θα πρέπει να δούμε την προχρηματοδότηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή να δούμε ένα καταποκοπήν ποσό που θα πρέπει να παρασχεθεί στα ΜΜΕ, στους βασικούς επιχειρηματίες. Άρα η Γενική Διεύθυνση για τις Υπηρεσίες εργάζεται για να εφαρμόσει μέτρα για την ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων σε όλους τους τομείς και τμήματα. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή πλατφόρμα η οποία να είναι ενιαία, η ερμηνεία θα πρέπει να είναι ενιαία καθώς και η εφαρμογή. Όλα αυτά βοηθούν για την μείωση της γραφειοκρατίας, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Καρβάλιο στην έκθεσή της. Η έκθεσή σας, κυρία Καρβάλιο, ήταν πραγματικά πολύτιμη για μένα και τις υπηρεσίες μου για να δούμε πού θα πρέπει να προωθήσουμε αλλαγές για να φτάσουμε σε μια πραγματική απλούστευση. Ως προς τη στρατηγική της Λισαβόνας, γιατί να θεωρήσουμε ότι η στρατηγική καινοτομία θα λειτουργήσει τη στιγμή που δεν λειτουργήσε η στρατηγική της Λισαβόνας. Στη στρατηγική της Λισαβόνας έχουμε μία στοχοθέτηση του 3%. Το κρατήσαμε αυτό και στην καινοτομία οι Υπουργοί Ερευνών το προώθησαν αυτό το ζήτημα καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς έτσι ώστε ο προϋπολογισμός για την έρευνα να υφίσταται πίεση σε όλα τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να δώσουν μάχη, μια πραγματική μάχη οι Υπουργοί Ερευνών έτσι ώστε να κρατήσουν τον υπάρχοντα προϋπολογισμό ή να τον επαυξήσουν. Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι ενώ η Ένωση της Καινοτομίας θα, θεωρώ ότι θα λειτουργήσει, η έρευνα και η καινοτομία είναι στο επίκεντρο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ετέθη από τον πρόεδρο Μπαρόζο. Η Επιτροπή θεώρησε ότι είναι το επίκεντρο η πεμπτουσία της πολιτικής μας και τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο πρόεδρος Βον Ρομπόη θα το συζητήσει σε μια ειδική διάσκεψη το Δεκέμβριο. Χρειαζόμαστε λοιπόν input από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για να είμαστε σίγουροι ώστε αυτό που έκανε η Φιλανδία όταν γνώρισε μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες στη δεκαετία του 90 έτσι ώστε να επενδύσει μέχρι και το τελευταίο ψυχείο που διέθετε στην έρευνα. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ευρύτερα, γιατί είδατε που οδηγήθηκε η Φιλανδία σήμερα με αυτή τη συνεισφορά. Θα πρέπει να πείσουμε τους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων λοιπόν να υποστηρίξουν την Ένωση της Καινοτομίας. Επίσης, εάν δούμε τους στόχους μας, τον στόχο 3% για έρευνα και ανάπτυξη και πολύ αναφερθήκατε και στο δίκτυ, οι δίκτες ε, καινοτομίας. Η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό τον ε, ε, καθηγητή Μάσκολει θεώρησα ότι θα πρέπει να μας δώσει όχι πληθώρα δικτών, αλλά έναν ενιαίο δίκτυ. Στο τέλος όμως μου ελέγχθη ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος δίκτυς ο οποίος να ενέχει όλα αυτά τα στοιχεία. Και συνεργαστήκαμε και με τον ΩΣΑ επί του θέματος αυτού. Γνωρίζω ότι δεν μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε έναν ενίο δείκτη. Δεν μπορεί ένας δείκτης να τα αποτιμήσει όλα. Οι ΙΠΑ εργάζονται για έναν ενιαίο δείκτη και το πάνελ υψηλού επίπεδου μου ανέφερε ότι χρειάζονται δύο χρόνια για να εργαστούμε για αυτόν τον ενιαίο δείκτη. Στο μεταξύ όμως δεν κρίναμε σκόπιμο απλώς να κρατήσουμε στάση αναμονής επί δύο χρόνια. Είδαμε λοιπόν αυτό το βαθμολόγιο καινοτομία. Έχουμε 25 δεδομένα, στο παράτημα 1 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Με συγχωρείτε, στο παράτημα 2 διορθώνει η Επίτροπος. Αν δούμε τους ανθρώπινους πόρους, τα επικερδή συστήματα έρευνας, τα links και την επιχειρηματικότητα, τα ε, διανοητικά περιουσιακά στοιχεία και ούτω καθεξής, θεωρούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία ακριβώς τα χρειαζόμαστε σε αυτό το σύνθετο, σε αυτό το σύνθετο βαθμολόγιο για να εμπεριέχει τα πάντα, δηλαδή να καλύπτει όλες τις οπτικές γωνίες και να μπορεί να ε, συγκρατεί όλες αυτές τις ε, πληροφορίες και να συγκρίνει τα συγκρίσιμα. Αυτά είναι τα ζητήματα που εφήγησαν από τα μέλη. Στην ακρόασή μου μου είπατε ότι υπερεύαινα το χρόνο μου. Αυτό, θέλετε, αυτό με πιέζετε νομίζω. Θέλετε να με πιέσετε για να μου επιστήσει την προσοχή σε αυτό και τώρα. Εν πάση περιπτώσει, προχωρούμε όχι μόνο υπό την ε, Ουγγρική Προεδρία. Ήδη συναντήθηκα με τον ε, Ούγγρο Υπουργό Έρευνας για θέματα καινοτομίας και είδαμε πώς ε, οι εταιρικές σχέσεις θα προωθηθούν υπό την Ουγγρική Προεδρία. Επίσης θα έχουμε την ενδιάμεση ε, αξιολόγηση μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας για να δούμε πώς θα προετοιμάσουμε το πρόγραμμα πλαίσιο, το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο, που θα, όπου θα εμπλακεί και η Ουγγρική Προεδρία και θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μία ε, πολιτική καινοτομίας η οποία βρίσκεται σε ένα ράφι και είναι στατική. Για να επιτηρήσουμε λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο χρειαζόμαστε τη δική σας συμμετοχή. Εγώ χρειάζομαι την άμεση υποστήριξή σας. Η Ένωση Καινοτομίας θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή μόνο όταν δράσουν από κοινού όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Αυτό είναι ύψης της σημασίας για την πολιτική μας. Έχουμε κοινωνικές ε, επιταγές που δεν μπορούν να λυθούν από μεμονωμένα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτές τις κοινωνικές ε, προκλήσεις. Χρειάζομαι την υποστήριξή σας για την ε, σύλληψη αυτή των εταιρικών οικονομικών σχέσεων στον τομέα της ε, καινοτομίας και ελπίζω να ε, δοθεί η άδη, δηλαδή το πράσινο φως, από το Συμβούλιο Υπουργών το Δεκέμβριο. Και όσο προχωρήσει το πιλωτικό εταιρικό σχέδιο και δούμε τι αποκομίζουμε, και τι διακυβέρνηση θα προωθήσουμε, όλα αυτά τα επιμέρους ε, ζητήματα θα συμβάλλουν στο σύνολο. Και ελπίζω να με υποστηρίξετε στεναρά για να προωθήσω αυτή την κοινοτική, κοινοτικά καθαρά πολιτική. Κυρία Επίτροπε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πληροφόρηση, για το χρόνο που μας διαθέσατε και νομίζω ότι έτσι προχωρήσαμε και εντός των επομένων εβδομάδων θα μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα στενά. Ευχαριστώ πολύ και θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξης. Ερχόμαστε λοιπόν στο επόμενο θέμα και όπως σας είπα έχουμε αναστρέψει το 5 και το 6 και έτσι ξεκινάμε με το παλιό 6 νυν 5 δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον Γενικό Προπολογισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδιατύπωση. Ο κύριος Κάλφιν έχει το λόγο σαν εισηγητής. Δεν είναι εδώ. Α, όχι, με συγχωρείτε, τώρα τον είδα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Θα σας παρουσιάσω μία πολύ αρχική γνωμοδότηση ε, για το θέμα μου διότι πολλά από τα ερωτήματα δεν έχουν ακόμη απαντηθεί και από πλευράς διαδικαστικής και όσον αφορά το περιεχόμενο του ε, δημοσιονομικού κανονισμού που όπως ξέρετε είναι η ραχοκοκαλιά του γενικού προϋπολογισμού και της διαδικασίας τους περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία, είναι οριζόντιος ε, και αναφέρεται εις, ε, τα, τις δαπάνες και στα έσοδα. Συνήθως κάθε τρία χρόνια εξετάζουμε αυτό το θέμα και τώρα πρέπει να κάνουμε τη δεύτερη αναδιατέπωση. Υπάρχει και μία αλλαγή στη διαδικασία και θα επανέλθω σε αυτό. Ουσιαστικό οι ιδέες του δημοσιονομικού κανονισμού είναι να χρησιμοποιήσουμε και να καταστήσουμε πιο απλό τον προϋπολογισμό, να τονίσουμε όλες τις, ε, ε, όλους τους πόρους και ε, να τονίσουμε επίσης την, τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στον τομέα αυτό. Προσπαθούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι στην εφαρμογή των δημοσιονομικών αρχών, να ε, δρομολογήσουμε τις ανταλλαγές με τους εταίρους μας, να βασιστούμε σε προγράμματα που να βασίζονται στην απόδοση και ε, σε συνολικά ποσά και σε μέθοδους ελέγχου. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Και από την άποψη της δικιάς μας Επιτροπής, αφού ακούσαμε την ε, Επίτροπο αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές ε, οι αρχές που ακούγονται πάρα πολύ ωραίες δεν ε, συνάδουν με τα προγράμματά μας και ουσιαστικά την χρηματοδότηση της έρευνας και θα τονίσω καταρχήν τις ε, τη διαδικασία διότι δεν έχουμε πλέον συμβουλευτική ε, διαδικασία αλλά συναπόφαση. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ πιο σαφή ρόλο στην ε, υιοθέτηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μία διαδικασία αναδιατύπωσης. Δηλαδή όλες οι προηγούμενες ε, τροπολογίες του ο προϋπολογισμού δεν μπορούν να αλλάξουν και αυτό δημιούργησε ερωτήματα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και η κυρία Γκρέσλε, η συγγήτρια, ζήτησε από την νομική υπηρεσία μία γνωμοδότηση για τη δυνατότητα να εξετάσει αυτή τη διαδικασία διότι έτσι περιορίζεται το Κοινοβούλιο ή στην εξέτασή του του εγγράφου, στη δυνατότητα της διατύπωσης τροπολογιών και αλλαγών. Ε, λοιπόν, Περιμένουμε ακόμη την τελική απόφαση της νομικής υπηρεσίας της κυρίας Γκρέσλε αλλά βάσει των διαβουλεύσεων που είχαμε μέχρι τούδε προτιμά να ε, επιστρέψει την, στην Επιτροπή την πρόταση και να ξεκινήσουμε με μία νέα πρόταση οπότε θα έχουμε ε, πλήρη δυνατότητα να τροποποιήσουμε το κείμενο που μας προτείνουν. Βέβαια θα δούμε τι θα αποφασίσει η Επιτροπή Προϋπολογισμού που ηγείται σε αυτή τη διαδικασία και αν αποφασίσουν ε, να επιστρέψουμε θα, θα περιμένουμε με τις προτάσεις μας για την ε, αναδιατυπωμένη μορφή η οποία θα εξεταστεί από το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, δηλαδή το περιεχόμενο του δημοσιονομικού κανονισμού, θέλω να αναφέρω ορισμένα στοιχεία, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικά για την Επιτροπή μας και διευκολύνομαι από την εξαιρετική παρουσίαση και, τον, και τη συζήτηση με την Επίτροπο διότι η πρόταση της Επιτροπής ΙΤΡ είναι ότι έχουμε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα ε, στην χρηματοδότηση της καινοτομίας στον προϋπολογισμό και Έχουμε τα σχόλια της κυρίας Καρβάλιο και ε, πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε και να δρομολογήσουμε τις καινοτομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, ο δημοσιονομικός κανονισμός πρέπει να βρει μια ισορροπία μεταξύ ε, της ευελιξίας και της ε, υποχρεώσεως αποδόσεως λογαριασμών. Και από αυτού θέλω να ε, ζητήσω ορισμένες διευκρινήσεις, διότι ένα από τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός αποβλέπει εις την αποφυγή κινδύνου και εις ε, την μηδενική κινητοποίηση. Πράγμα το οποίο ε, ε, καλό είναι για να χρηματοδοτεί κανείς τα τρέχοντα αλλά στην καινοτομία εάν δεν έχουμε και δεν αναλαμβάνουμε κανένα κίνδυνο δεν μπορεί να υπάρξει υποκίνηση για καινοτομία. Όσον αφορά την πρόσβαση εις ε, τη χρηματοδρότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους μεμονωμένους ερευνητές, πρέπει να υπάρξει μία απλοποίηση των διαδικασιών που να τονιστεί όταν θα διατυπώσουμε προτάσεις και ένα άλλο θέμα είναι η διατήρηση της ε, δημοσιονομικής ε, πειθαρχίας χωρίς όμως ε, να αυξάνουμε τους κινδύνους και ε, υπάρχουν πολλά κείμενα τα οποία θα πρέπει να επανεξετάσουμε προτού υιοθετήσουμε το, την τελική μορφή του κειμένου. Στην έκθεση της κυρίας Καρβάλιο που αναφέρεται επίσης στο δημοσιονομικό κανονισμό με την αύξηση των ποσών και της χρηματοδοτήσεως ενός συγκεκριμένου ποσού είναι πράγματα τα οποία ε, νομίζω ότι μας παραπέμπουν στην έκθεση Καρβάλιο για να ζητήσουμε ένα νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Ε, ξέρω βέβαια ότι το Συμβούλιο δεν πολύ ε, ενθουσιάζεται αλλά εμείς θέλουμε να υπάρξει καινοτομία στα προγράμματα. Το Συμβούλιο δεν θέλει να ξαναδημιουργεί, να ξαναχρησιμοποιεί ε, τα ε, ποσά τα οποία ε, κερδίζονται αντί να τα επιστρέφει στα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε όμως ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ καλά τέτοια διαθέσιμα για την χρηματοδότηση της καινοτομίας. Προηγουμένως μιλήσαμε για το ανεκτό επίπεδο κινδύνου το οποίο αναφέρεται στο αποδεκτό ποσοστό κινδύνου ιδίως όσον αφορά τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας και υπάρχει μία κοινή, ε, ένα κοινό θέμα ε, ότι δηλαδή ε, πρέπει να υπάρχει ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Δεν θα επισέλθω σε άλλες λεπτομέρειες ε, όσον αφορά το συγκεκριμένο κείμενο του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό θα γίνει σε περίπτωση όπου η Επιτροπή που ηγείται ε, συνεχίσει να επεξεργάσει το κείμενο αντί να ε, επιστρέψει με ένα νέο. Γι' αυτό και θα δούμε αναλόγως των εξελίξεων αν θα συνεχίσουμε κατευθείαν με την αξιολόγηση του δημοσιονομικού κανονισμού ή αν θα περιμένουμε έως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, παρουσίασε ένα νέο κείμενο για να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Άλλος ζητά το λόγο ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός φάκελος αυτός γιατί αποτελεί την βάση για οτιδήποτε άλλο θέλουμε μετά, παραδείγματος χάρη στο πρόγραμμα πλαίσιο 8, εάν δεν υπάρχει δημοσιονομικός κανονισμός, δεν ε, μπορούμε να κάνουμε τίποτα στο πλαίσιο στο πρόγραμμα πλαίσιο. Είναι η βάση λοιπόν για οτιδήποτε θέλουμε, για το αν θα πραγματοποιηθεί ή όχι. Νομίζω πως ένα από τα βασικά ζητήματα, και θα το δούμε στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης, είναι η αξιολόγηση αντικτύπου. Να δούμε δηλαδή ποιος θα είναι αυτός ο έλεγχος και όλες αυτές οι διατάξεις και τι σημαίνουν αυτά για τους ε, ενδιαφερόμενους όχι αυτούς οι οποίοι κάνουν τον έλεγχο ή εκδίδουν κανονισμούς, αλλά κυρίως για αυτούς οι οποίοι υφίστανται αυτές τις διατάξεις και γνωρίζουμε πως τα ερευνητικά προγράμματα πολύ συχνά είναι η δαπάνη πολύ μεγαλύτερη από το όφελος τη στήριξη που λαμβάνει δηλαδή κανείς. Νομίζω πως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι πολύ απλά το ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση αντικτύπου οπωσδήποτε για τις μικρομισές επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν να υπογράψουν συμβάσεις 30 ε, ή 50 σελίδων και μετά να ακολουθούν 500 σελίδες υποσημειώσεων και όλα αυτά βέβαια να μην αντιστοιχούν καθόλου με την ενίσχυση την οποία λαμβάνουν. Πρέπει λοιπόν να γίνεται, όπως σας είπα, αυτή η αξιολόγηση αντικτύπου από την πλευρά των ενδιαφερομένων που ενισχύονται και όχι μόνο από την πλευρά της διοίκησης. Να υπάρχει δηλαδή και μία αναλογικότητα εδώ πέρα. Και υπάρχουν κάποιες δυνατότητες εξοικονόμησης. Όλοι ξέρουμε τις προτάσεις από το One Stop Shop μέχρι το ένα ενιαίο έντυπο για όλους για να έχουμε και γρήγορες και αποτελεσματικές προθεσμίες πληρωμών, αλλά αυτά θα γίνουν μόνο εάν αποκτήσουμε τώρα τον δημοσιονομικό οργανισμό. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος, ε, ο Ντί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μέσα στα πλαίσια της τριετούς αναθεώρησης του βασικού κανονισμού θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για αυτή την διεξοδική εργασία. Πρόκειται για καινοτομίες πολύ σημαντικές που λαμβάνουν υπόψη τα νέα στοιχεία ως προς τις δημόσιες προμήθειες και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μελετήσουμε. Αυτός ο δημοσιονομικός κανονισμός εισαγάγει την καινοτομία ότι μπορούν να ε, γίνουν να δανειοδοτήσεις μέσα στα πλαίσια των ευρωομολόγων όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής, αλλά μόνο για τα ακίνητα. Στον δημοσιονομικό κανονισμό, σε σχέση με τις ε, μεγάλες ε, επενδύσεις, με στα πλαίσια των μεγάλων επενδύσεων, έχουμε μεγάλες δυσκολίες να εισαγάγουμε πολύετής συναλλαγές που υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές προοπτικές. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο μπορούμε να εισαγάγουμε ε, τροπολογίες για να μην προβλέπεται αυτή η τριετής αναθεώρηση και να έχουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο έτσι ώστε να ε, στοιχειοθετήσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε καθαρά λογιστικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Κανένας άλλος δεν ζητάει το λόγο, οπότε για σήμερα τελειώνουμε με αυτό το σημείο της μέσης και Περνάμε στο σημείο 6 για καλύτερη ρύθμιση δηλαδή, το είχαμε ήδη συζητήσει αυτό και τον λόγο έχει ο κύριος Τσίτσεστερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή είναι μια γνωμοδότηση ανεξάρτητων ε, εκτιμήσεων και μπορώ να σας πω ότι βρεθήκαμε ως σκιώδη στην ε, προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο και έτσι καταφέραμε να φτάσουμε σε έξι τροπολογίες συμβασμού σε σχέση με ορισμένα από τα σημεία που έφυξαν οι συνάδελφοι. Δεν φτάσαμε σε ομοφωνία, δυστυχώς. Άρα θα πρέπει να ψηφίσουμε ορισμένες τροπολογίες ξεχωριστά. Επειδή οι συνάδελφοι με τους οποίους ε, συζήτησα τη τροπολογίας συμβασμού δεν, επειδή οι συνάδελφοι αυτοί δεν είναι παρόντες, είναι κάπως δύσκολο να μπούμε σε λεπτομέρειες. Δεν θα ήταν σκόπιμο να γίνει κάτι τέτοιο. Χαίρομαι για τη συνεργασία που επετεύχθη με την κυρία Ριέρα Μαντουρέλ και με τους φίλους μου στο ΕΛΚ για τα περισσότερα ζητήματα. πέρα από αυτό το θέμα, αν θέλετε μπορούμε να δούμε τις τροπολογίες σε λεπτομέρεια, αλλά θα ήταν άκερο αν λάβουμε υπόψη την αθρώα παρουσία των συναδέλφων εδώ. Ίσως ο κύριος Ρούμπιχ ε, έχει ορισμένα σχόλια και θα, θα τα περιμένω για να απαντήσω. Δεν έχω μπροστά μου το κείμενο των τροπολογιών συμβιβασμού, αλλά τις ε, ετοιμάσαμε και συμφωνήσαμε. Γι' αυτό ε, ελπίζω να μπορέσετε να ε, διανύμετε τις τροπολογίες ή σήμερα ή αύριο το πρωί. Πάντως συμφωνήθηκαν σε επίπεδο σκιωδών. Παουλ Ρουμπίχ έχει τον λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τζάιλς Τσίτσεστερ. Νομίζω πως οι 7 συμβαστικές τροπολογίες με τον ε, κύριο Μπένσεν, τον σχεδιοδησίτη, νομίζω ε, είναι κάτι που μπορούμε να υποστηρίξουμε και ο ΣΕΛΚΑ. Τρία σημεία είναι για εμάς σημαντικά. Πρώτον, ανεξάρτητοι έλεγκτες, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τους αξιολογήσει και όχι οι υπάλληλοι της Κομισιόν και βεβαίως να υπάρχει διαφάνεια στην ε, νομοθεσία αυτή και όσον αφορά, όπως σας είπα, τους ενδιαφερομένους ε, οι οποίοι θα πρέπει να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν μετά τις ε, συνέπειες. Επίσης για την εξελόγηση επιπτώσεων της νομοθεσίας ειδικά όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, όχι μόνο το κόστος, αλλά το τι σημαίνει στον διεθνή ανταγωνισμό αυτό για τις επιχειρήσεις. Πρέπει να μπορούν να διασφαλίσουν θέσεις εργασίας στον διεθνή ανταγωνισμό οι επιχειρήσεις μας, οπότε θα πρέπει να γίνεται αυτή η ανεξάρτητη αξιολόγηση, είναι ιδιαίτερο σημαντική και βεβαίως αυτό αφορά πολύ περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες φτάνουν πολύ γρήγορα στα όρια τους όταν μιλάμε για το κόστος και να μπορέσουν βεβαίως να έχουν και επαρκές ε, και επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό και αυτό επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά τους. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω και αυτό είναι το τρίτο θέμα που μας απασχόλησε με τις ε, αλλαγές ε, στην προστασία των μητέρων και τις υποχρεωτικέ άδειε πατρότητας. Εκεί πέρα δεν είχαμε επαρκή αξιολόγηση αντικτύπου. Δεν ξέραμε ε, τι σημαίνει αυτό το οποίο ψηφίζουμε στο Κοινοβούλιο και το τι θα πρέπει να κάνουν ε, οι επιχειρήσεις και στις 27 χώρες και οι ενδιαφερόμενοι. Αν ξέραμε λοιπόν τι γίνεται και με τις ε, θέσεις εργασίας και με τη χρηματοδότηση, ενδιαφέρον θα ήταν ε, και για το τμήμα εδώ πέρα της ε, έρευνας πολιτικής να μας πει τι αντίκτυπο θα έχει. Για να δούμε βεβαίω πώ θα το συμβάσουμε και την Ατζέντα 2020. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Τσίτσιστερ και νομίζω πω ήταν πολύ καλή η εκθεσή του. Ευχαριστώ και εγώ για αυτά τα οποία είπατε. Είναι κρίμα το ότι... Ναι, σας είδα. Ε, το ότι δεν είναι πολύ περισσότεροι συνάδελφοι εδώ πέρα. Γιατί αυτό είναι από τα βασικά προβλήματά μας. Πρέπει να το πω ως πρόεδρος. Βασικό πρόβλημα στην πολιτική και νομοθετική μας εργασία ότι είτε σπάνια είτε καθόλου όταν ε, λαμβάνουμε τις πολιτικές αποφάσεις δεν γίνεται κάποια έρευνα και δεν ασχολούμαστε και εμείς με τις συνέπειες προσπάθησα με νομοθετικές ε, πράξεις να μπει στην ημερήσια διάταξη η αξιολόγηση αντικτύπου. Και θα ήμουν ευγνώμων να συνεχιστεί αυτό στο μέλλον. Αλλά και να το συζητήσουμε, γιατί τότε έχει νόημα η συζήτηση να ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες των πράξεων μας. Και θα ήθελα να προσθέσω πως ε, πέραν αυτών των οποίων πρότεινε η Κομισιόν θα πρέπει να κάνουμε και μία αξιολόγηση αντικτύπου για τις α, ε, ιδέες ε, τις οποίες έχουμε εδώ πέρα και εισάγονται από το Κοινοβούλιο, γιατί καμιά φορά ακούγονται εδώ πέρα κάποιες έξιμες ή όχι τόσο έξιμες προτάσεις και δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει κάτι, αλλά το αποφασίζουμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έχουμε εδώ πέρα στην πρόταση και θα έπρεπε νομίζω και στην άλλη να ασχοληθούμε λίγο. Παρακαλώ και ο συνάδελφος εκεί στο βάθος θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα τον λόγο εξ ονόματος της κυρίας Τερέζα Ριέρα η οποία ακόμα έχει προβλήματα μεταφορών αλλά μου ζήτησε βεβαίως να πω την αποψή της για την γήτρια από το Μάσο Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τον κύριο Τσίτσεστερ, ε, όπως ε, πάντα, όπως λέει συνάδελφος, για την καλή συνεργασία. Έχουμε νομίζω φτάσει σε μια συνεργασία με την οποία θα διατηρήσει το δικαίωμα πρωτοβουλίας η Κομισιόν, αλλά θα μπορέσουμε έτσι να έχουμε μια αξιολόγηση αντικτύπων από τους ειδικού για να αυξηθεί η ποιότητα της νομοθεσίας. Επίσης έχουμε τη συμβαστική τροπολογία 2 με την οποία υπερασπίζουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Βεβαίως οι οικονομικές στοιχείες δεν μπορούν να προηγηθούν των ε, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, εδαφικών ε, πτυχών και των πτυχών της δημοσιογία και βεβαίως ε, της, της μεγαλύτερης ελπίζουμε πως οι περισσότερες ομάδες θα υποστηρίξουν την θέση μας για την ε, δημοσίευση του σχεδίου αξιολόγηση που πριν φτάσουμε στη νο... νομοθετική πρόταση. Σας ευχαριστώ. Τζάιλς, έχετε πάλι τον λόγο. Uh, ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και την ε, επικοδομητική τους αντιμετώπιση. αποτολμώ να πω ότι λείπουν τόσα πολλά ε, μέλη επειδή κατά βάθο εμπιστεύονται τον ε, εισηγητή. Αυτό θα το δούμε βέβαια αύριο κατά την ψηφοφορία. Ελπίζω η κυρία Ριέρα Μαντουρέλ να είναι ευτυχής με τις προτάσεις συμβιβασμού. Δεν έχουμε ακόμα επιβεβαίωση, αλλά ίσως εσείς έχετε περισσότερες πληροφορίες από μένα. Θα ήθελα να σταθώ στο εξής βασικό σημείο που ανέφερε και ο Πόλο Ρούμπιχ. Πολύ συχνά πρέπει να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια χωρίς να έχουμε πλήρη γνώση των γεγονότων. Και βεβαίως πολλές φορές ε, βασιζόμαστε σε συναδέλφους άλλων επιτροπών για να καλύψουν ε, αυτά τα ζητήματα. Αλλά τα σχόλιά του σε σχέση με την άδεια μητρότητας που δημιουργεί μεγάλη ανησυχία στο δικό μου κράτος ως προς το ε, ενεχόμενο κόστος, σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν μελέτες αντικτύπου και η εξαιρετική αυτή εργασία μπορεί να προωθηθεί μόνο αν γίνει μια ανεξάρτητη μελέτη αντικτύπου. Ελπίζω λοιπόν οι συνάδελφοι να με υποστηρίξουν αύριο το πρωί κατά την ψηφοφορία χωρίς ε, μεγάλες δυσκολίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστεί και ο Πρόεδρος και νομίζω... Ε, ε, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε για τις συμβασικές τοπολογίες, οπότε αύριο θα μπορέσουμε να το ψηφίσουμε Οπότε ολοκληρώθηκε η μερίσια διάταξη. Μπορούμε να, μπορεί να λήξει η συνεδρίαση, αλλά σε μερικά λεπτά όταν θα είναι εδώ όλοι οι συντονιστές θα μπορέσουν να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν όλοι παρίστανται ήδη. Ευχαριστώ.